Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά θέματα για σήμερα και έτσι κι αλλιώς και αυτό από χθε, το 2015. Έχουμε την ειδική έκθεση του ε, Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ότμπο, να μας παρουσιάσει αυτή την ειδική έκθεση πριν δώσω το λόγο στον συγητή μας. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο και ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Έχετε ήδη ορισμένα πράγματα για την, για την έκθεση παρακολούθησης, οπότε θα είμαι σύντομος. Πολύ Ε, χρειάζεται η παρακολούθηση. Η ειδική έκθεση είναι η πρώτη γενεά της ε, έκθεσης παρακολούθηση. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο έχει σκοπό να προβεί σε αυτή την παρακολούθηση μέσω έκθεσης κάθε χρόνο στο μέλλον. Αυτή τη φορά είχαμε, 5, είχαμε 7 ειδικέ εκθέσεις και θα σας πω τι διαπιστώσαμε. Ότι η Επιτροπή έχει ένα εύρυθμα λειτουργών σύστημα σε σχέση με την παρακολούθηση των συστάσεων ε, του ελεκτικού συνεδρίου και των ετοιμάτων της ε, ε, αρχής προϋπολογισμού και βλέπουμε ότι υπάρχει συμμόρφωση με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής. Είδαμε επίσης ότι υπήρχαν κάποια περιθώρια βελτιώσεων στο σύστημα της Επιτροπής. Θα ήθελα, όπως και εχθές, να ε, επιστήσω την προσοχή του ε, εισηγητή, φαντάζομαι θα το είδε ήδη, ότι η παρακολούθηση του ελεγκτικού συνεδρίου έχει να κάνει με τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Θέλαμε να συμπεριλάβουμε και το αίτημα του Κοινοβουλίου, αλλά δεν το κάναμε. Και θα ήθελα να... Ε, σας ρωτήσω αν θέλετε από τις εκθέσεις της δικές σας παρακολούθησης να μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε στο μέλλον ε, στην εκθεσή μας, όπως επίσης και τις, τα αντίστοιχα αιτήματα του Συμβουλίου. 70% των συστάσεων ε, που ε, συμπεριλήφθηκαν στις 7 εκθέσεις ε, έχουν εφαρμοστεί σχεδόν πλήρως. Είμαστε ικανοποιημένοι με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένω γωνίο σε συνεργασία με την Επιτροπή για στο μέλλον για πιο διεξοδικές εκθέσεις παρακολούθησης. Θα αρκεστώ σε αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, κύριε Πρόεδρε και ε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μέλη της ε, Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τα σύντομα εισαγωγικά σας σχόλια. Και θα ήθελα τώρα να δώσω ε, σύντομα τον λόγο προς τον εισηγητή μας, τον κύριο Γκάια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Όπ για την παρουσίασή του και θα είμαι πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, το θετικό ε, συμπέρασμα είναι ότι η Κομισιόν ένα ε, μεγάλο κομμάτι των συστάσεων του ηλεκτρικού συνεδρίου το λαμβάνει υπόψη και το εφαρμόζει. Και εμείς ε, με μεγάλη μας χαρά να δούμε κατά πόσον ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το πώς είναι οργανωμένο το σύστημα αυτό στην Κομισιόν, κατά πόσον το σύστημα αυτό εξυπηρετεί ή όχι. Καθότι ε, το 70% εφαρμογή σημαίνει ότι το 30% δεν εφαρμόζεται. Άρα δηλαδή υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Αλλά καταρχήν τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά όπως και η σύσταση για το LIFE. Αυτή η σύσταση δεν αγνοείται πλήρως από την Κομισιόν και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να επανέλθουμε στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για τη δουλειά του και εκεί που απευθύνεστε στην ε, Επιτροπή θέλω να πω ότι εγώ ως εισηγητής αρμόδιος για την απαλλαγή θέλω να σχολιάσω το εξής. Εάν θέλετε, βεβαίως θα ήταν χρήσιμο στις απόψεις να λάβετε υπόψεις και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί καθαρά θεωρητικά είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε διαφορετικά εμείς ε, μία θέση του ελεγκτικού συνεδρίου ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας πούμε, όταν επρόκειτο για το leader, πολλοί από εμάς, ε, λόγω της ε, εμπειρίας τους από την Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία επίσης ασχολήθηκε με το ε, πρόγραμμα Leader. Εμείς λοιπόν δεν ακολουθήσαμε όλες τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ανεξάρτητος ε, θεσμός. Ε, συνεργαζόμαστε με μεγάλο, μεγάλη χαρά για, στις εισηγήσεις σας, εκθέσεις αλλά πιστεύω ότι η πλειοψηφία των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου τελικά ε, γίνεται αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πλειοψηφία αυτών των ε, προτάσεων εγκρίνεται από την Ολομέλεια. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι συμπίπτουν οι απόψεις μας σε όλα τα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήταν χρήσιμο ή πολύ φιλικό αν θέλετε το να λάβετε υπόψη σας την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όσον αφορά τις απόψεις του ελεγκτικού συνεδρίου για ε, την ε, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ αυτές τις απόψεις θα τις λάβω υπόψη μου, διότι μία έκθεση ε, follow-up για το follow-up, για το follow-up, για τη συνέχεια, είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή και πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστεί. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι ως Επιτροπή Προϋπολογισμών να δούμε πώς ακριβώς εξετάζουμε τις εκθέσεις ε, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, στο επίπεδο των συντονιστών εδώ και αρκετό καιρό θα με το θέμα αυτό. Η πρώτη μας ιδέα ήταν να καταρτίζουμε κανονικές εκθέσεις και μετά αυτό το εφαρμόσαμε σε πάρα πολλέ ειδικέ εκθέσει. Η κυρία Αντρέαισεν για την Ελία, ο κύριο Ντότ για ένα θέμα που τώρα δεν το θυμάμαι όμω, ο κύριο Μαρινέσκου ε, πρόσφατα για την ε, ε, πάυση λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων, για τον παροπλισμό τους και ε, επειδή λοιπόν είχαμε αυτό το προηγούμενο των τριών εκθέσεων, διαπιστώσαμε ότι οι ιστορικές υπηρεσίες ε, του κάθε οργάνου έχουν διαφορετική άποψη για το πώς συντάσσονται οι εκθέσεις. Ας πούμε, οι εκθέσεις Αντρέασεν και Ντόιτς ε, ήταν στην ημερήσια ε, διάταξη για την Ολομελία και μετά αφαιρέθηκαν διότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου θεώρησαν ότι αυτές δεν είναι κανονικές εκθέσεις όπως προβλέπει ο κανονισμός. Έκτοτε λοιπόν έχουμε μια εσωτερική συζήτηση με τα όργανα του Κοινοβουλίου για το τι ακριβώς θα κάνουμε με τις ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει πλήρης ομοφωνία στους συντονιστές ως προς το ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιλαμβάνεται με τα συμπεράσματα του συνεδρίου στο σύνολό του. Και όχι μόνο ως Επιτροπή Προϋπολογισμών, γιατί αυτά που λέτε δεν αφορούν μόνο εμάς, αλλά και άλλες επιτροπές. Και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα γίνει αυτό. Έχοντας λοιπόν κατά νου ότι εμείς ε, δεν μπορούμε να συντάξουμε κανονικές εκθέσεις. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Η μία είναι να ανακαλύψουμε νέα μορφή εκθέσεων. Αυτό ε, καθαρά συστηματικά είναι η πιο καθαρή μέθοδος, όμως ε, θα διαρκέσει και η άλλη δυνατότητα που έχουμε ως συντονιστές είναι να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει σήμερα ο κανονισμός να προάγουμε αυτές τις εκθέσεις στην Ολομέλεια ως προτάσεις πρωτοβουλίας, ως προφορικές προτάσεις προς την Κομισιόν ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Αυτό το επιλέγουμε εμείς. Νομίζω βέβαια ότι αυτή δεν ενδείχνεται ως μέθοδος για όλες τις εκθέσεις. Και επειδή όπως σας είπα πρόκειται για το follow-up του follow-up της Κομισιόν, η έκθεση ότι είναι πολύ σημαντική και θέλω να τη λάβω υπόψη μου στην απαλλαγή, αλλά σας λέω για καμία από τις άλλες δυνατότητες ε, που ε, προσφέρει ο κανονισμός ε, δεν θα έλεγα το ίδιο. Κατόπιν τούτου προτείνω στους συναδέλφους να επανέλθουμε στην πεπατημένη βέβαια η πεπατημένη σημαίνει ότι θα καταρτήσω, θα συστήσω συντάξω ένα έγγραφο και αυτό θα είναι αντικείμενο της απαλλαγής. Εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι το θέμα αυτό θα το λάβω υπόψη μου στην απαλλαγή και ε, θα σας το αναφέρω όταν θα εξετάσουμε ε, την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, τον κύριο Γκάια που είναι ο εισηγητής. Ε, δεν βλέπω να υπάρχουν ε, άλλοι που να ζήσαν το λόγο. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Οπ κατά πόσο επιθυμεί να τοποθετηθεί σε αυτά που είπε ο κύριος Γκάια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα πολύ επικοδομητικά του σχόλια και θα ήθελα απλώ να προσθέσω ορισμένα πράγματα που και που όταν το ελεγκτικό συνέδριο προβαίνει σε μια δεύτερη ειδική έκθεση που καλύπτει ένα θέμα το οποίο έχει καλυφθεί και προηγουμένως, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα σχόλια και οι συστάσεις θα ληφθούν υπόψη και στην ε, δεύτερη έκθεση. Από ό,τι κατάλαβα, ζητάτε από το ελεγκτικό συνέδριο να λάβει υπόψη και τα αιτήματα του Συμβουλίου αλλά και του Κοινοβουλίου ε, στις ε, εκθέσεις παρακολούθησης στο μέλλον. Από ό,τι κατάλαβα, επίσης τονίσατε και κάποια παραδείγματα για τα οποία θα μπορούσε να υπάρχει διάσταση απόψεων σε σχέση με την κατεύθυνση των συστάσεων ε, μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και κοινοβουλίου δηλαδή να συμπεριληφθούν και αυτά σε μια μελλοντική ειδική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τον εισηγητή. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω και την Κομισιόν να τοποθετηθεί ο κύριος Κραφ θα πάρα πολύ σύντομο, ε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτό το νέο είδο ηθική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου γιατί δίνει μια περιεκτική αξιολόγηση των συστάσεων, ε, της παρακολούθησης των συστάσεων. Τα θετικά σχόλια που λάβαμε σε σχέση με την εφαρμογή ε, τα λαμβάνουμε υπόψη, αλλά λαμβάνουμε υπόψη βέβαια και τι αδυναμίε, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί γιατί κάποιε διαδικασίε παρακολούθηση θα δώσουν τη δυνατότητα σε υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να έχουν μια έγκαιρη, γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση, όχι μόνο στα συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και στα αιτήματα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και θα γνωρίζετε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια ανακοίνωση ε, και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την παρακολούθηση των συστάσεων που, ελήφ, που ε, υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ορίζει απαλλαγής. Ευχαριστούμε πολύ και εσά, κύριε Κράφτ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα και ευχαριστώ όλους τους μετέχοντες γιατί κάπως τώρα παραμένουμε πιστοί στο χρονοδιάγραμμά μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον η Γενική Γραμματέας έχει ήδη έρθει. Μήπως είναι εδώ. Ήρθε. Πολύ ωραία. Παρακαλώ να την ενημερώσετε. Ε, μέχρι τότε πάμε ε, στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμόν 12. Πρόκειται για την απαλλαγή του 2011, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τμήμα 3 Επιτροπή. Και ε, για το θέμα αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο να καλωσορίσω καταρχήν την κυρία Κάθριν Ντέι, την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Ντέι, σας καλωσορίζουμε στη συνεδρίασή μας. Βεβαίως ε, είσαστε πάντα προσκεκλημένοι ε, στην Επιτροπή μας. Αν θέλετε μπορείτε προφανώς να καθίσετε εκεί. Ε, φέτος ο συγκητής μας είναι ο κύριος Γκάια από τους Σοσιαλιστές. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουμε τα μέλη ΟΠ και Μουκουρούσα. Θα ήθελα να ζω τον εισηγητή κατά πόσον επιθυμεί ε, να λάβει το λόγο ή αν πρέπει να ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό, το Ελεγκτικό Συνέδριο. κύριος Γκάια. Θα ήθελα λοιπόν ε, να απευθυντώ στη Γενική Γραμματέα πρώτα απ' όλα. Και κυρία ε, Ντέι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Εσείς έχετε ένα πολύ δυσάρεστο καθήκον. Δηλαδή, Ό,τι δεν θέλουμε να συζητήσουμε με τους επιτρόπους, τα λέμε σε εσά. Και αυτό θα προκύψει και σήμερα από τις ερωτήσεις. Αυτές που ετέθησαν μέχρι τώρα σε εσά είναι γενικής φύσεως. Σήμερα θέλω να αναφερθώ σε ένα ειδικό θέμα, να το συζητήσουμε μαζί. Πρόκειται για την έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή λοιπόν η έκθεση προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τι είναι αυτή η έκθεση αξιολόγησης. Τα λέω έτσι πολύ προσεκτικά, ψάχνω τα βλόγια μου. Ε, είναι ένα είδος performance audit, ένα είδος ε, αξιολόγησης απόδοσης. Αυτό που αξιολογούμε είναι κατά πόσον ε, εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Τώρα βέβαια τίθεται το θέμα κατά πόσον αυτό είναι επίκαιρο ή όχι. Είμαι ευγνώμων στην κυρία Μακόσκα από τη Γραμματεία, η οποία, ε, κυρία Μακόσκα, ως μία από τους τρεις αρμόδιους, με βοηθάει να συντάξω την ε, έκθεση απαλλαγής. Αυτή λοιπόν η κυρία Μακόσκα μου την εξή πληροφορία. Το ε, Αμερικανικό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει το 90% των περιπτώσεων μόνο κάτω από το πρίσμα της απόδοσης και όχι της ε, συμβατότητας, της compliance. Τίθεται λοιπόν, τώρα το πω κάπως ηρωνικά, το εξής ερώτημα. Αν μία γέφυρα έχει ε, κατασκευαστεί σωστά και τη χρησιμοποιούν όλοι, πάβει να έχει ενδιαφέρον το σε ποια ακριβώ χρονική στιγμή κατατέθηκαν τα χαρτιά συμμετοχή στο διαγωνισμό, αν κατατέθηκαν πέντε λεπτά νωρίτερα ή όχι από την καταληκτική ημερομηνία. Τι θέλω να πω, ότι ε, τα λάθη ε, και πόση σημασία έχουν τα λάθη και τα σκάνδαλα. Ε, καλό αυτό να το συζητάμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε περισσότερο την ουσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την άποψή μου, δικαίως και σωστά έχει πρόβλημα με αυτή την έκθεση αξιολόγησης. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό των 130 εκατομμυρίων ευρώ με κοινή διαχείριση. Και μιλάμε για χιλιάδες προγράμματα Άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταρτήσει μια ικανοποιητική έκθεση που να μην είναι τεράστια σε όγκο να είναι εύχριστη και ευσύνοπτη. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα καθήκον που το καθήκον αυτό αναγκάζει σχεδόν και καταδικάζει την Επιτροπή να αποτύχει. Πάντα θα βρίσκουμε κάτι που δεν θα μας αρέσει, ότι δεν θα είναι αρκετά εκτενής, δεν είναι αρκετά ακριβής, εξετάζει λάθος παραμέτρους. Η Κομισιόν λοιπόν, σας είπα, είναι καταδικασμένη να κάνει λάθος. Και αυτό δεν είναι ευχάριστο. Εγώ τώρα, κοιτάξτε, φιλικά τα λέω όλα αυτά, με φιλική διάθεση. Οι δύο συνάδελφοι πρώοι μου που ασχολήθηκαν με την απαλλαγή και την έκθεση αξιολόγησης ήταν πολύ καυστικοί. Για μένα όμως ακόμα αυτό το θέμα δεν είναι καθοριστική σημασίας γιατί κατανοώ ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει αυτό το δυσεπίλητο πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν και με τις υπηρεσίες της Κομισιόν αλλά και με άλλους συναδέλφους στην πολιτική μου ομάδα να ξεκινήσουμε συζήτηση να δούμε μα τι περιμένουμε από αυτήν την έκθεση και πώς μπορούμε να την ε, φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μικρή σε όγκο, να έχει πολιτική σημασία και από αυτήν να προκύπτουν συμπεράσματα που να βοηθάνε την Κομισιόν. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Το μόνο που μου ήρθε κατά νου είναι το εξής. Σε αυτή την ε, έκθεση Και πριν από την σύνταξη της έκθεσης πρέπει να έχουμε διάλογο με την κυρία Κάτριν Ντέι και με τους ε, συναδέλφους της. Και να δούμε γιατί να μην το συσχετίσουμε αυτό με την Ευρώπη 2020. Να πούμε ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία για την ευρωπαϊκή πολιτική η οποία ευτυχώς συνοδεύεται και από στόχους. και να πούμε ότι εμείς ως ελεγκτές είμαστε ικανοποιημένοι αν η Κομισιόν λαμβάνει τα σωστά μέτρα για να επιτύχει τους στόχους της. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι το εξής. Να μας εξηγήσει η Κομισιόν τι ρόλο παίζουν οι εμβληματικές πρωτοβουλίες. Η κακομήρα Κομισιόν, και το κακομήρα δεν το λέω ηρωνικά, το εννοώ. Η κακομήρα λοιπόν η Κομισιόν δέχεται επιθέσεις διότι οι προσδοκίες που συνδέονται με αυτή την έκθεση δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Άρα δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε πολιτικά τι περιμένουμε από αυτήν την έκθεση αξιολόγησης. Και αφού συμφωνήσουμε μετά να διατυπώσουμε έναν κατάλογο προσδοκιών, να απευθύνουμε τον κατάλογο αυτό στην Επιτροπή και πάνω σε αυτά τα κριτήρια να κρίνονται στο μέλλον οι εκθέσεις αξιολόγησης. Εγώ θέλω να δουλέψω πάνω σε αυτές τις παραδοχές. Βεβαίως ε, και θα κάνω σχόλια, αλλά νομίζω δεν θα ήταν δίκαιο ε, να ζητάμε τώρα από την Κομισιόν μία έκθεση αξιολόγησης με βάση κριτήρια τα οποία όμως δεν μπορεί, στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Πρέπει να δούμε πρώτον αν μπορούμε να δουλέψουμε με την έκθεση αυτή και δεύτερον αν μπορούμε να εξάγουμε λογικά πολιτικά συμπεράσματα. Και τρίτον, αν δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, να δούμε κατά πόσον επικρίνουμε τους πραγματικά υπέτειους. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ πιο επικοδημοτικό από το να λέμε κάθε χρόνο στην Κομισιόν φέρτε μας του χρόνου δύο κιλά περισσότερο χαρτί που όλοι ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι πόσο δύσκολο είναι να τα επεξεργαστεί κανείς όλα αυτά και να καταλήξει μια επικοδομητική εργασία. Αυτά είχα να πω σήμερα το απόγευμα αλλά βέβαια δεν θέλω να εμποδίσω κανένα συνάδελφο να υποβάλει συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν ξέρω, θέλετε και οι δύο το λόγο ή υπάρχει κάποιος που επιθυμεί να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Επιτροπή ήδη συζήτησε το ζήτημα των δαπανών των υπολείπων θεσμικών οργάνων και τώρα εξετάζουμε τα ευρήματα που αφορούν τα δαπάνες της Κομισιόν που αποτελούν το 67% των συνολικών διοικητικών δαπανών όλων των κοινωνικών οργάνων τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που έκανα στι τελευταίες μου παρεμβάσεις στο σημείο 2 της Μεσής Διατάξεως ε, μπορούν πλήρως να εφαρμοστούν στο κεφάλαιο 9 αυτής της έκθεσης, έκθεσης στο Ελληνικό Συνέδριο καταλήγει ότι οι διοικητικές δαπάνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάστηκαν από από τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Τώρα, σε σχέση με την Κομισιόν, διαπιστώσαμε κάποιες αδυναμίες σε δύο τομεί. Μία αφορά στον υπολογισμό πληρωμέ κοινωνικών επιδομάτων προς τους υπαλλήλους και το δεύτερο αφορά την διαδικασία προμηθειών. Σε 15 από 18 περιπτώσεις οι πληροφορίες για την προσωπική και κοινή κατάσταση των μελών των υπαλλήλων θεωρήσαμε ότι δεν ήταν σαφής σχετικά με τις προμήθειες διαπιστώσαμε κάποιες αδυναμίες σε τρεις περιπτώσεις κατά την εφαρμογή των κριτηρίων μας στην διαδικασία επιλογής και κάποιες ε, ασυνέπειες ε, ε, στην διαδικασία αυτές. Επίσης, σε ό,τι φορά τα, τις συμβάσεις, ένας από τους υποβάλλοντες δεν αποκλείστηκε σύμφωνα με τα κριτήρια περί εμπειρίας Πρόεδρε, θα αναφέρω ότι οι συστάσεις που έκανε το όργανό μας προς όλα τα θεσμικά όργανα αφορούν και στην Κομισιόν σχετικά με την προσωπική κατάσταση του προσωπικού και τις διαδικασίες προμήθειας. Μπορώ να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής. Το άρθρο 319 προβλέπει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια έκθεση αξιολόγησης και αυτή η έκθεση θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι της ε, διαδικασίας απαλλαγής. Η έκθεση Κομισιόν ε, του Φεβρουαρίου του 2012 ε, έλαβε απάντηση τον Ιούνιο του 2012 και η έκθεση που έφτασε τον Νοέμβριο απαντήθηκε μέσω επιστολής ε, από εμάς. Σε ό,τι φορά την πρώτη έκθεση αξιολόγησης, το συνέδριο κατέληξε ότι αυτή η έκθεση ήταν αδύναμη και είχε πολύ λίγη αξία. Η δεύτερη, έκθεση αξιολόγηση ε, αποτέλεσε μια σημαντική πρόοδο και η Κομισιόν τα σε όλους ε, τους τομείς δραστηριοτήτων και πολιτική. και το διαπιστώσαμε και δηλώνει για μια κομφορά ότι ήταν μια σαφής πρόοδος. Η Κομισιόν επίσης εκτίμησε ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω τα πράγματα, κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Διότι το δεύτερο μήνυμα το οποίο συνήγαγα από την έκθεση εξελόγησης δεν παρήχε αξιόπιστες, αξιόπιστα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Και ο εισηγητής νομίζω πώς αναφέρθηκε στην συμφωνία ανάμεσα στην Κομισιόν και το Συνέδριο σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει και πώς θα πρέπει να προχωρήσουν από εδώ και στο εξή. Το Ελεκτικό Συνέδριο, σε ό,τι αφορά το μέλλον, είπε ότι χρειάζεται ένα αξιόπιστο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων που θα επιτρέψει την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Και δεύτερον, αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει με την υποβολή της ε, αίτησης αυτής, ε, έκθεσης αυτής αξιολόγησης. Μία σειρά αποδράσεων, αποδράσεις θα πρέπει να αναλάβει η Κομισιόν και εμείς συστήσαμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για την διαχείριση και το σύστημα υποβολής εκθέσεων που θα αφορά την ε, <clears throat> διαδικασία υποβολής της έκθεσης αυτής της, στα όργανα απαλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Όπο. Ακούσαμε το ελεκτικό συνέδριο και θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω την κυρία Ντέι να μιλήσει εξ ονόματος Κομισιόν. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας, να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι και πάλι που ξανάρθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ετήσια πρόσκλησή σας ε, <clears throat> ως ε, ε, τμήμα της διαδικασίας απαλλαγής να παρευρεθώ. Το Νοέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη της έκθεση σε σχέση με τα αποτελέσματα που πέτυχε και είναι σύμφωνα με το άρθρο 318 της ε, ε, συνθήκης. Έχουμε λάβουν υπόψη τις ενδείξεις και από το Γινοβούλιο και από το Ελεκτικό Συνέδριο στην πρώτη έκθεση. Άκουσα πολύ προσεκτικά ε, όλα αυτά που είπε πέρσι η Επιτροπή σας και λάβαμε υπόψη τα σχόλια και την κριτική σας στη δεύτερη έκθεση. Κατά την άποψή ε, και χαίρομαι ε, όλος ιδιαίτερος ε, που ακούω αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου. Πιστεύουμε ότι αυτή η δεύτερη έκθεση έχει μια πιο περιεκτική προσέγγιση. Επίσης χαίρομαι που οι βελτιώσεις ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη έκθεση λαμβάνονται υπόψη και στις γραπτές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής σας, στις οποίες απαντήσαμε νωρίτερα μέσα αυτή την εβδομάδα. Τη δεύτερη έκθεση τώρα παρέχει αξιολόγηση για όλες, όλους τους τίτλους προπολογισμού για να φύγουμε από αυτή την επιλεκτική προσέγγιση που είχαμε στην πρώτη έκθεση, οπότε τώρα έχετε μια περιεκτική προσέγγιση που πιστεύω ότι συνάδει με ε, τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου. Εντοπίζει βασικούς τομείς ε, ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, αποτελεσματικότητας, ε, και δείχνει ότι ε, τα κονδύλια ανταποκρίνονται στους στόχους των προγραμμάτων. Και αυτό ε, που νομίζω ότι είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό και ενδεικτικός προς την αξία της έκθεσης είναι ότι βλέπουμε διάφορες μεταβολές στην απόδοση. Ξέρουμε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο εκπνέει, είναι η τελευταία χρονιά φέτος του τρέχοντος πλαισίου, οπότε μπορούμε να κάνουμε ακόμη μία ενδιάμεση μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαια ακόμη πολύ ε, σίγουροι ε, σε σχέση με τα αποτελέσματα όλων των προγραμμάτων, Παρόλα αυτά ε, υπάρχουν ήδη κάποια διδάγματα, έχουν γίνει κάποιες προσαρμογές ε, είτε στα τρέχοντα προγράμματα ή στα, στα προγράμματα στα οποία ε, μαθαίνοντας από τα λάθη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει αλλαγές στον επόμενο γύρο προγραμμάτων. Τούτων λεχθέντων είμαστε οι πρώτοι που βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και θέλουμε να, βελτιώσουμε, να συζητήσουμε ενδεχόμενες περαιτέρω βελτιώσεις. Σε σχέση με αυτά που είπε το ελεγκτικό συνέδριο μόλι ε, συμφωνούμε ε, σε μεγάλο βαθμό με αυτά που αναφέρει το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχέση με το πού πρέπει να ε, συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και τους στόχους μας. Βελτιώνουμε το εσωτερικό μας σύστημα για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων για την επόμενη χρονιά, για τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς και βάσει του νέου πλαισίου που θα μας πάει μέχρι το 2020. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέσα, ε, δηλώσεις δραστηριοτήτων, ετήσιες δηλώσεις, αξιολόγηση και ε, τους ε, ελέγχους επιδόσεων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρέπει να βρούμε μια σωστή, ένα σωστό συνδυασμό input και να παρακολουθούμε ολόκληρη τη διαδικασία για να έχουμε πραγματικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και προστιθέμενη αξία. Όπως επίσης και για να έχουμε καλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία μας. Πρέπει να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό. Βασιζόμαστε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να διατηρήσουν το απλούστερο πλαίσιο πλαίσιο που πρότεινε για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε ένα ισχυρό ε, ε, πλαίσιο παρακολούθησης. Έχω κάποιες ανησυχίες γιατί όταν βλέπω πόσο περίπλοκα ξαναγίνονται τα πράγματα με τις διαπραγματεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή βλέπω κάποια απώλεια απλότητας ε, και σαφήνειας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω έκκληση και σε εσά και στο Συμβούλιο να μας βοηθήσουν να είμαστε απλούστεροι ε, και σε ένα, σε ένα πλούστερο σύστημα το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε πιο εύκολα στο μέλλον. Ετοιμαζόμαστε ήδη για την επόμενη έκθεση αξιολόγηση, θα καλύπτω 2012. Το ελεκτικό συνέδριο ζήτησε να δημοσιευθεί πολύ νωρίτερα, οπότε προσπαθούμε προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε την επόμενη έκδοση της έκθεσης με την έκθεση σύνθεσης ε, για τις δραστηριότητες διαχείρισης που κανονικά τον Ιούνιο δημοσιεύουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα καλύψουμε μόνο επιπλέον μερικούς μήνες, αλλά είναι καλύτερα από το τίποτα. Ε, νομίζω δηλαδή ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο αρμονικά και κάθε χρόνο να ε, παράγουμε αποτελέσματα που θα είναι πιο χρήσιμα για τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος ε, κύρια Ντέι. Τώρα άρχεται η συζήτηση. Ευχαριστούμε για τα ουσιαστικά σχόλια. Σας είχαμε στείλει γραπτές ερωτήσεις, λάβουμε και γραπτές απαντήσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους της ε, Επιτροπής. Η πρώτη που έχει δει το λόγο είναι η συντονίστρια του ΕΛΚ, η κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γενική και γραμματέα που ήρθατε και πάλι κοντά μας. Ε, πολύ ενδιαφέρον το να μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Ξεκινώ λοιπόν με ένα πρόβλημα που με εντυπωσιάζει όχι μόνο εμένα αλλά και τους ε, συναδέλφους. Τουλάχιστον υπήρξαν κάποιοι που μου το ανέφεραν. Ο τρόπος με τον οποίο αποκτάμε τις πληροφορίε ε, Έχει φτάσει η στιγμή Μάλλον, από τότε που είπατε ότι οι απαντήσεις ε, δεν πρέπει να είναι πάνω από 25 ε, γραμμές, ε, όλο και λιγότερο απαντάει η Κομισιόν. Και ρωτώ, γιατί το είπατε αυτό. Εγώ υποβάλλω γραπτές ερωτήσεις και νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αν οι ερωτήσεις απαντώνται όπως είναι το σωστό έτσι ώστε να προκύψει κάποια ουσιαστική απάντηση. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο εάν τα παραρτήματα για τις ε, γραπτές ερωτήσεις μπορούσαν να διατεθούν σε όλους. Γιατί ε, κάνουμε την εξή εμπειρία. Τα παραρτήματα ε, υποβάλλονται μόνο στους ενδιαφερόμενους ευρωβουλευτές και όλοι οι άλλοι αρχίζουν να ρωτάνε. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να μπορούμε να έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό. Αυτό τώρα που λέω έχει σχέση με την περίπτωση Νταλή. Ο Γενικός ε, Διευθυντής ε, της Όλαφ έδωσε στα μέσα ενημέρωσης περισσότερες πληροφορίες από ό,τι στο Κοινοβούλιο. Και όταν ρωτήσαμε, μα γιατί έγινε αυτό και ε, λίγο πολύ είπε ότι η Κομισιόν, συγκεκριμένη αυτή η περίπτωση, η Γενική Γραμματεία διέγραψε στοιχεία από την απάντησή του. Ε, το είδαμε αυτό και πέρυσι ε, στο ε, καταστατικό, όταν γίνεται το λόγος για το καταστατικό, διαψώσαμε το ίδιο. Το βρίσκω λοιπόν ιδιαίτερα λυπηρό. Και το ερώτημα που τίπτε είναι πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, δεν θέλω να μακρηγορήσω κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλω κάποιες πληροφορίες. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Τουλάχιστον τα ερωτήματα που θέτουμε τώρα να απαντώνται στην ε, ερώτηση 44, όπου τι το ερώτημα, πόσες θέσεις καλύπτονται με διαγωνισμούς και πόσες χωρίς αυτούς. Η απάντηση δεν δίδεται, είναι ακρεμή. Επίσης, θα με ενδιέφερε ε, θα σας τα πω ότι δεν έχει απαντηθεί. Θα φτιάξω έναν κατάλογο και ίσως σε ένα δεύτερο γύρο μπορούν να απαντηθούν όλα αυτά. Δεν το βρίσκω σωστό οι ερωτήσεις που υπεβάλλουμε να μην απαντώνται ή τόσο πρόχειρα έτσι ώστε να είναι άχρηστη η απάντηση. Αυτά στο θέμα απάντηση και μη απάντηση. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, ερώτηση 53 όπου πρόκειται για την κινητικότητα των γενικών γραμματέων. Θέλω να γνωρίζω πόσοι γενικοί διευθυντές μέχρι τώρα έχουν ε, επηρεαστεί από αυτή την κινητικότητα. Γιατί από ό,τι φαίνεται εσείς ε, δεν χρειάζεται να υφίσταστε τη γεννητικότητα, την κινητικότητα, ενώ όλοι οι άλλοι την υφίστανται και μάλιστα εξαναγκάζονται και προς αυτή. Παραδείγματο χάρη, ο κύριος Ρέκλιν, ο Γενικός Γραμματέας ε, του ΕΚΟΦΗΝ, είπε ότι δεν δέχεται την μετάθεση και μετά τον απολύσανε. Να δούμε λοιπόν κατά πόσον οι κανόνες ισχύουν για όλους ή για τους περισσότερους μόνο. Αυτοί οι κανόνες για τους περισσότερους. Εδώ ε, ο επαναδιορισμός ε, του Μισελ Πετίτ ως Προέδρου της ε, Ad Hoc Επιτροπής για τη Διοντολογία. Πρέπει, και το είπα αυτό στον κύριο Μπαρόζο, ότι είναι λυπηρό για την αξιοπιστία της Κομισιόν ότι κάποιος ο οποίος έρχεται από την Κομισιόν έχει μία υπέρογγη σύνταξη, πάει μετά σε ένα δικηγορικό γραφείο και εντάσσεται σε μία ομάδα λόμπι. Αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα λυπηρό. Τελικά θεωρώ ότι ισχύει αυτό που λέμε σε ελληνικά μεταφρασμένο έγινε από δήμαρχος κλητήρας και αυτό το βρίσκω προσβολή για τον κύριο αυτό. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ε, προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε σχετικά με το ε, σύστημα της ε, εκπεριτροπής κάλυψης θέσεων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ υπάρχουν κάποιες προποθέσεις ε, και είναι δεσμευτικό αυτό το σύστημα με ορισμένους όρους βέβαια όπως η ηλικία. Και αν ερμηνεύω σωστά τους όρους ισχύει αυτό που σας είπα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το εκπεριτροπή σύστημα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως σε σχέση με την εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη προς τα έξω. Νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά την ε, εκπεριτροπής μετακίνηση των ε, γενικών διευθυντών, εμείς είμαστε υπέρ αυτού γιατί είναι ένα θέμα ε, που έχει σχέση με τη διαφάνεια, με την δημοκρατική νομιμοποίηση και δεν καταλαβαίνω γιατί προβλέπονται εξαιρέσει. Αυτές οι εξαιρέσει πώς αιτιολογούνται. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω ίσως πώς μπορεί κανείς ε, να αιτιολογήσει αυτές τις αλλαγές. Αν θέλει κάποιος να ξανά αποκτήσει ένα γενικό γραμματέα, τότε γιατί δεν συμπεριλαμβάνετε στην αξιολόγηση μια ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για να νομιμοποιήσετε αυτή την κίνηση. Αν θέλετε λοιπόν τη δημοκρατική νομιμοποίηση, τότε γιατί συμπεριλαμβάνετε και περισσότερους σε αυτήν. Αλλά τώρα δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό που κάνετε. Προβλέπετε εξαιρέσει εσεί ε, και ξέρετε ε, τι έχει συμβεί με αυτές τις εξαιρέσεις. Έχουμε προκαλέσει δυσπιστία και γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε να μας δώσετε ε, σαφείς ε, πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα τη μέθοδο αξιολόγησης. Εδώ ομολογώ ότι η Κομισιόν έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά καθήκοντα. Συνάδελφε Γκάιρα, αυτό που προτείνατε εσείς το βρίσκω τη χειρότερη λύση. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν συμφωνούμε. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε τους δίκτες που ισχύουν στην στρατηγική 2020, όπως αριθμός των αποφύτων ε, λυκείων ή αριθμός των παιδιών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ε, ερωτώ λοιπόν, εμείς ε, οι Ευρωπαίοι για τέτοιου είδου πράγματα φέρουμε ευθύνη. Ας πούμε, το σχολικό σύστημα στην Βόρεια Νέα Βεσφαλία ή στην Ελλάδα, αν αυτό πάρει η Κομισιόν, ποιο τιμωρειται ουτε η κομισιον ουτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οι ντόπιοι επιτόπου έχουν πρόβλημα. Να πάρουμε τώρα τους δείκτες της στρατηγικής 2020 για να ξεκινήσουμε την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προϊστάμενης αξίας, εγώ δεν συμφωνώ. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω και αυτό να το λάβει υπόψη της η Κομισιόν, η ίδια η Κομισιόν να δει που έχει αρμοδιότητες. Μόνο εκεί μπορεί κανείς ε, να ε, υπολογίσει την προσθέμενη αξία και όχι έτσι στο πολύ φλού τι είναι η κοινωνική Ευρώπη. Ή στο θέμα των υποδομών. Τι κατασκευάστηκε, που βοηθήσαμε, που δώσαμε ανθρωπιστική βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια, ερευνητικά προγράμματα. Όλα δηλαδή εκείνα από τα οποία προκύπτει ευρωπαϊκή προστεμένη αξία και όχι όλα τα άλλα όπου δεν είμαστε ουσιαστικά αρμόδιοι. Αυτό το βρίσκω επικίνδυνο το να περιλαμβάνουμε και όλα αυτά στην αξιολόγηση. Συνοψίζοντας λοιπόν θέλω να πω το πρώτο ερώτημά μου αφορά το εκπεριτροπή σύστημα, το δεύτερο αφορά τη μέθοδο αξιολόγησης. Ο συνάλφος κ. Γκάια κατέθεσε μία πρόταση, κατέθεσα κι εγώ και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας δώσει έτσι γενικά, μας δώσει γενικά ε, ε, απόψεις, θεωρίες για το τι είναι η ευρωπαϊκή προστιμένη αξία. Όχι γενικά όμως, δεν θέλουμε γενικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Πώς ακριβώς μπορούμε να επιτύχουμε ευρωπαϊκή προστιμένη αξία. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ο κύριος Μπαλτσίτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν βέβαια διάφορα ευρωπαϊκά γραφεία και υπάρχουν και διάφορα συμφέροντα. Αυτό το θέμα νομίζω ότι πρέπει να αναλυθεί και ενδεχομένως και να πρέπει να αλλάξουν κάποιες δομές για να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Εσείς πιστεύετε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι ικανοποιητική ή μήπως ε, θα πρέπει να αλλάξουν οι αρχές έτσι ώστε όλα ε, τα εξωτερικά γραφεία να λειτουργούν με βάση τους ίδιους κανόνες και να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ντέ, κυρία Ντέ, εδώ, εδώ είμαι. Απέναντί σας, αλλά έδρα της Προεδρίας. Σας καλωσορίζω και να θέσω μια ερώτηση σχετικά με την οδηγία περί καπνού, την υπόθεση Νταλή. Επανειλημμένα διαβάσαμε πως η διαβούλευση η υπηρεσιακή για την οδηγία περί του καπνού δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται σε ένα γράμμα του ε, Ιανουαρίου. Η κυρία Τεστόρη έκανε διάφορες παρατηρήσεις ε, και αναφέρθηκε ότι δεδομένου ότι το ζήτημα είναι πολύ ευαίσθητο από πολιτική σκοπιάς. δεν ε, θεωρώ πως μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την ενδοϊπηρεσιακή συνεννόηση και διαβούλευση. 156 ε, ερωτήσεις υπολήθηκαν, κάποιες υπηρεσίε ε, απάντησαν σε ορισμένες εξ αυτών, όπου αναφέρεται σε μία ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέχρι τον Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Και σε εξηγώ το γιατί δεν, χρειάζεται, δεν μπορούμε να τροποποιούμε το χρονοδιάγραμμα ε, το γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά αυτές οι διαβουλεύσεις ενδοϊπηρεσιακές νομίζω είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να καταργούμε την παρουσίαση μιας πρότασης, την υποβολή μιας πρότασης. Έχει συμβεί και στο παρελθόν για μια ενδοϊπηρεσιακή διαβούλευση, δηλαδή να καταργηθεί αναμένοντας ε, την ε, συνεδρίαση μιας ολομέλειας του Κοινοβουλίου ή ενός ε, Συμβουλίου. Τον Οκτώβριο μιλούσαμε στο Συμβούλιο για την κρίση του ευρώ και σίγουρα όχι για την οδηγία περί καπνού. Τώρα, σε ό,τι φορά διαφάνεια, αυτό για το οποίο επικρίνεται ο κύριος Νταγή, ο πρόεδρος Μπαρόζο τον επικρίνει ότι παραβίασε κάποιους κανόνες ε, του ΠΟΕ σε θέματα καπνού. Υπάρχουν πάλι όμως της ε, Κομισιόν που είχαν επαφές με διαφόρους ε, εμπλεκόμενους στην υπόθεση του καπνού. Είναι συνήθις πρακτική υπάλληλοι εκτός της υπηρεσίας ΣΑΝΚΟ, της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, διότι αυτή είναι που ασχολείται με το θέμα. Ποια είναι και έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα που άπτουν του καπνού. Ήθιστε λοιπόν να γίνονται παρόμοιε συνεννοήσει εκτό τη νομική υπηρεσία των Κομισιών. Είναι φυσιολογικό λοιπόν άλλοι υπάλληλοι τη Γενική Γραμματεία ε, να έρχονται σε επαφή πριν από την ολοκλήρωση και την πραγματοποίηση τη ενδοπηρεσιακή ε, συνεννόηση και διαβούλευση, τώρα σχετικά με τι συναντήσει ε, τώρα στην ερώτηση 17 ε, στο κείμενο που περιέχει 160 περίπου ερωτήσεις αναφέρεται πως ε, έχετε καταγράψει τις επαφές που είχαν οι υπάλληλοι με τους ε, καπνοπαραγωγούς και μας αναφέρεται ότι με κάποιες εξαιρέσεις ο Γενικός Γραμματέας η νομική υπηρεσία δεν είχαν επαφές με τους μεγάλους διανομής. Αυτό είναι ένα ζήτημα σαφέστατο και παρά τότε και παρά τα αυτά ένα mail ε, απεστάλλει 17 και το ένα απόγευμα 17 και 10 σε κάποιον της Swedish Match αναφέροντας ότι ο κύριος Νταλή ε, παρετήθηκε μετά από την προσφυγή που είχε υποβληθεί το Μάιο 2012. Γιατί λοιπόν αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επαφών. Είναι, πρόκειται για επαφή μεταξύ ε, της υπηρεσίας σας ή ε, μόνο προσωπικά με τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες ε, για τον καπνό. Και σας θέτω το ερώτημα. Σας ενημέρωσαν για τα παράπονα που είχαν εκφραστεί και που αφορούσαν στην οδηγία περί καπνού. Και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ παράδοξο κύριε Αντέη σας ε, λένε πολλές φορές ότι είστε 28η επίτροπος, είστε η υψηλότερα ιστάμενη ισταμενη υπαλληλος Δεν θα έπρεπε να φροντίζετε οι προσφυγές ε, να ακολουθούνται από πράξεις. Είναι συνήθις πρακτική αυτή. Αυτό έχει πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν. Τώρα για τον κύριο Πετή ε, θα ερώτημα από την κυρία Κρέσλερ. Δεν θα επανέλθω, αλλά έχω μια ερώτηση σχετικά με τις συμφωνίες για τον καπνό. Η πρώτη συμφωνία ε, το 2004 συνήθι με τη Φίλιπ Μόρις, είχα συμμετάσχει και η ερώτησή μου είναι η εξή. Με δεν ε, θεωρείται ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στην υπόθεση περί καπνού που είναι και τόσο διάφανες ε, τώρα και τα, αν τα ευρωπαϊκά όργανα επιλέγουν κάτι το οποίο δεν συμφέρει την βιομηχανία καπνού μπορούν να καταργηθούν, έχουν γίνει παρόμοιες ε, πράξεις, ε, παρόμοιες αλλαγές και είχαμε συνάντηση με τον κύριο Σέρκοβιτς εδώ τον Νοέμβριο του 2012. Αυτή η συνάντηση αφορούσε τις ομάδες εργασίας των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται ε, για την Κομισιόν που κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Κομισιόν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο κ. Σέρκοβιτς το δήλωσε ο ίδιος. Θα θέλαμε να μας πείτε όμως τι γίνεται με αυτά τα προγράμματα για την τροποποίηση αυτών των ομάδων εμπειρογνωμών. Θα μπορούσατε να μας δώσετε επίση κάποια σχόλια για αυτά που διαβάζουμε στον τύπο ότι η ομάδα ψηλού επίπεδου του κ. Στόιμπλε, το οποίο συναντήσαμε εδώ πριν από μερικού μήνε και που ασχολείται με τα διοικητικά σήμερα. Διαβάζουμε λοιπόν στον τύπο, ο κύριο Στόιμπλερ χρησιμοποίησε αυτήν την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και να προσκαλέσει εμπειρογνώμονες μιας επιχείρησης ε, προκειμένου να κάνουν σχόλια για την οδηγία περί καπνού. Είναι, αυτές οι φήμες είναι σωστές, είναι αληθινές και είναι αποδεκτό μια ομάδα αρμόδια για την μείωση της γραφειοκρατίας να, ε, να εκφράζει άποψη για αυτό το ζήτημα. Υπήρξε παραβίαση των κανόνων, ναι ή όχι. Παρακαλώ να μου απαντήσετε. Derek Vaughan. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του γενικού προϋπολογισμού. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ε, ε, και συγκεκριμένα τον ε, προπολογισμό της Επιτροπής. Έχουμε κάθε χρόνο μεγάλη μάχη, τσακωνόμαστε με το Συμβούλιο για τις πληρωμές ε, και είδα ότι αυξήθηκαν οι δεσμεύσεις, αλλά συχνά δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν θέλουν να καταβάλουν τα ποσά και στο τέλος του χρόνου βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές, αρκετά κονδύλια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει. Ίσως κάποιες νομικές συμφωνίες τότε να μην ε, γίνονται σεβαστές και υπάρχει επίσης και το ενδεχόμενο θέμα να πρέπει να πληρώσει επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω των ε, καθυστερημένων πληρωμών. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες οικονομικές συνέπειες λόγω της έλλειψης καταβολών πληρωμών από προηγούμενα έτη αλλά και για το 2012. Θα γνωρίζετε ότι θέλουμε μείωση του 5% στο προσωπικό. Αυτό είναι ένα στόχο, φιλόδοξο στόχο, 5% κάθε 5 χρόνια. Ποια ανάλυση, τι ανάλυση όμω έχετε κάνει σε σχέση με το θέμα αυτό και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στα ε, θεσμικά όργανα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τη, το επόμενο θέμα που απασχολεί και εμάς και εσάς, θέλουμε να ευθυγραμμίζεται ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θέλουμε και εμείς να έχουμε μια καλή σχέση κόστους και ωφέλους. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω θα ήθελα να μας πείτε ε, πόσο κοστίζει η απάντηση στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών κάθε χρόνο το κόστος δηλαδή των ερωτήσεων που σας, επι... που σας ε, ε, θέτει η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών, πόσο στοιχίζει, αν έχετε κάνει μία ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βόγαν. Ο κύριος Λιμπεράτσκι είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε. ερωτήσω τον κύριο Στάις και τον κύριο Μπαλτσίτης. Κυρία ε, Ντέι, υπάρχει ένα θέμα το οποίο βάλατε στην άκρη, δηλαδή για την ε, τροποποίηση του πλαισίου που διέπει τι συγκρούσεις συμφερόντων. Εδώ και αρκετό καιρό διαρωτώμεθα ποια είναι τα διδάγματα που μπόρεσε να συνάγει η Κομισιόν μετά από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις συγκρούσεις ε, συμφερόντων ε, των οργάνων και των υπηρεσιών της Ένωσης. Ε, ε ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρόμοιες σχέσεις στο παρελθόν και πως ε, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σας πιστέψουμε, πιστέψουμε. Αν μας λέτε πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων τότε δεν θα υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει και αν έχουμε πρόβλημα βλέπουμε τι συμβαίνει. Ο Επίτροπος Νταλή χρειάστηκε να πληρώσει το τίμημα ο ίδιος προσωπικά. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση εκ μέρου ε, ε, τη ομάδα των φιλελευθέρων. Ο συνάδελφο κύριο Στά ανέφερε την ομάδα υψηλού επίπεδου, η οποία ασχολείται με το θέμα του διοικητικού άχθου. Και υπάρχει μία περίπτωση την οποία έπτυξε. Εγώ λοιπόν θα ήθελα έτσι γενικότερα να αναφερθώ σε αυτή την ομάδα υψηλού Στις γραπτές απαντήσεις, στις γραπτές μας ερωτήσεις δηλώνεται ότι η διαδικασία για την εξάντε εξέταση του γραφειοκρατικού κόστους είναι πολύ καλύτερα να γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να γίνει από ένα εξωτερικό γραφείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει τελικά με την ομάδα υψηλού επίπεδου ε, η οποία είναι αρμόδια για τον περισμό της γραφειοκρατίας μετά το 2014 θα επανέλθει ή γιατί πιστεύετε ότι μια εσωτερική αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι καλύτερη από το να γίνει η εξέταση αυτή από έναν τελείως ανεξάρτητο οργανισμό. Ίσως μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Από ό,τι βλέπω, η Επιτροπή δεν έχει να υποβάλει άλλες ερωτήσεις. Κατόπιν τούτου, κυρία Κάθριν Ντέι, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Για το θέμα των ε, ερωτήσεων του Κοινοβουλίου, θυμάμαι καλά, λαμβάνω πάνω από 2.000 το χρόνο 12.000, ε, κάτι το οποίο σημαίνει πολλή ανάλυση, πολλή δουλειά, πολλές μεταφράσεις ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι δεν έχει κανένα ανάλυση κόστους, νομίζω το Κοινοβούλιο το έχει κάνει ε, και είχαμε έρθει σε επαφή για το πώς είναι δυνατόν να απαντάμε σε ερωτήσεις αλλά να μειώνουμε το κόστος τη διαδικασία αυτή. Συχνά παίρνουμε ερωτήσει που αφορούν πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες δημοσίως. Μπορούμε να δώσουμε πολύ σύντομες απαντήσεις. Παρακαλούμε βρείτε στην τάδε ε, ιστοσελίδα ή στο τάδε, στην τάδε δημοσίευση τις ε, απαντήσεις σε αυτό που επιθυμείτε. Μπορούμε επίσης να δούμε κατηγοριοποίηση μέσω περιφερειών, διορθωτικά ταμεία κλπ. Να τους λέμε να μας στέλνει αναπεριφέρεια ή αναταμείο αντί ανα χώρα μέλος και έτσι μπορούμε και να είμαστε ταχύτεροι στη δουλειά μας και να δίνουμε όλες τις, ε, ερωτή να δίνουμε όλες τις απαντήσεις ερωτήσεις. Επίσης έχουμε βάλει και ένα όριο στους χαρακτήρες γιατί βλέπαμε ότι οι συνάδελφοι έγραφαν πάρα πολύ μακροσκελείς απαντήσεις, κάτι που δεν απαντούσε υποχρεωτικά στην ερώτηση. Δηλαδή επαναλάμβαναν την ερώτηση και μετά την απαντούσαν. Γι' αυτό βάλαμε τον περιορισμό ως χαρακτήρες. Θέλουμε λοιπόν να δίνουμε τις πληροφορίες που μας ζητούν, αλλά με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Συγγνώμη κυρία Γκρέσλε αν δεν λάβατε το, την απάντησή μας. Εμείς πάντως τη στείλαμε Απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις και την 44. Μπορώ να σας δώσω και, μια να σας δώσω και ένα αντίτυπο τώρα, αλλά πας περιπτώσει τις αποστήλαμε γέρος τις απαντήσεις μας. Συγγνώμη αν δεν τις λάβατε. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα Τη κινητικότητα υψηλόπαθμων στελεχών, ε, η κινητικότητα είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Εγώ είχα πολύ στην ε, σταδιοδρομία μου και μου είναι πάρα πολύ χρήσιμο το γεγονό ότι τώρα ω Γενικό Γραμματέα έχω δουλέψει σε τόσο διαφορετικά τμήματα τη Επιτροπή. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή μου τη γνώση. Όμω το Σώμα των Επιτρόπων αποφασίζει πώ γίνονται οι διορισμοί, πού ανατίθενται ε, οι διάφοροι συνάδελφοι. Ε, έχουμε κάποιου κανόνε, αλλά έχουμε ε, και κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν και κάποιες εξαιρέσεις. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα της αξιολόγησης, ε, ναι, είναι τεράστιο εγχείρημα, πράγματι. Θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω, ε, για μας να προσπαθήσουμε να αποφασίσουμε με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια τι θέλουμε να επιτύχουμε με τις εκθέσεις σε βάση του άρθρου 318. Γιατί το να παρακολουθούμε τις στόχους ε, του, της στρατηγικής 2020 είναι πολύ ευρύτερο θέμα από την παρακολούθηση των στόχων για την εφαρμογή και την απόδοση των ε, ε, προγραμμάτων ε, από τα οποία, των προγραμμάτων που καλύπτονται από τα διάφορα ταμεία. Είδαμε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να στοχεύουν περισσότερο προς την στρατηγική 2020. Αυτό όμως μένει ακόμη να αποφασιστεί και πρέπει να δούμε με τα κράτη-μέλη πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Θέλουμε καταρχάς να έχουμε τη νομική βάση και το πλαίσιο και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να ορίσουμε ένα σύστημα παρακολούθησης κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει σύν το χρόνο να, παρουσια... να παρακολουθούμε πόσο επιτυγχάνουμε τους στόχους αυτούς. Αλλά ο προπολογισμό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τον προπολογισμό που διατίθεται σε εθνικό επίπεδο στου τομεί που καλύπτονται από του στόχου αυτού. Θέλουμε πάντοτε λοιπόν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν μπορούμε από μόνοι μα να κάνουμε μια σημαντική διαφορά, αλλά ελπίζουμε να είμαστε καταλήτη για να μπορέσει να κινηθεί η πολιτική προ τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το θέμα των ε, υπηρεσιών. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι αποκινούμε το Κοινοβούλιο ε, περάσαμε πολύ χρόνο να δούμε πώς ε, διαρθρώνονται αυτές οι υπηρεσίες και φτάσαμε πέρσι σε μία συμφωνία μεταξύ Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να προσπαθήσουμε σταδιακά να αναδιαμορφώσουμε, να δούμε όλες τις ε, υπηρεσίες πώς λειτουργούν, να αναδιοργανώσουμε εκείνες των οποίων οι δομές δεν είναι πλέον οι κατάλληλες κατά τη γνώμη μας. Θέλουμε όχι εναρμονισμένη βέβαια προσέγγιση για κάθε υπηρεσία, αλλά κάποιε κοινέ αρχέ. Α πούμε, σε μερικέ υπηρεσίε δεν εκπροσωπείται καθόλου η Επιτροπή, σε άλλα είναι πολύ μεγάλο το Διοικητικό Συμβούλιο και ούτω καθεξή. Προσπαθούμε να δούμε πώ θα το καταφέρουμε αυτό. Πέρσι στο τέλο τη χρονιά, εμεί δημοσιεύσαμε ένα χάρτη πορεία για να δούμε πώ θα κινηθούμε προοδευτικά προ αυτό το στόχο για τη βελτίωση δηλαδή τη δομή των υπηρεσιών. Θα ήθελα όμω να πω ότι η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη απευθεία για αυτό το θέμα. Μερικέ φορέ είναι τμήμα, συμμετέχει, παρακολουθεί τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν έχει από μόνη της την ευθύνη των υπηρεσιών αυτών. Είναι μια κοινή ευθύνη. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα με την οδηγία για τον ε, καπνό. Ε, θα ήταν, ε, είναι σημαντικό καταρχάς να πω ότι στο σημείωμα που συνυπέγραψα με τον γενικό γραμματέα της νομικής υπηρεσίας είπα, δεν είπα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαβούλευση, είπα ότι θα έπρεπε η έναρξή της να καθυστερήσει λίγο. Αυτό θα ήθελα λοιπόν να διορθωθεί. Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να γίνει, είπα ότι ίσως πρέπει να καθυστερήσει η έναρξή της. Εμεί, ε, στη Γενική Γραμματεία και στη Νομική Υπηρεσία κάνουμε την οριζόντια δουλειά μας, δηλαδή να εξασφαλίζουμε ότι οι προτάσεις τη επιτροπή ε, συμμορφώνονται με τους κανόνες που η Επιτροπή αποφάσισε. Θα μπορούσα να το συνοψίσω ως εξής. Έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίζουμε τη συνοχή της γενικότερης πολιτικής, ευρύτερης πολιτικής. Εμείς είμαστε αυτοί που εξασφαλίζουμε ότι η Επιτροπή σέβεται τη συμφωνία πλαίσιο ε, με το Κοινοβούλιο, ε, ότι ε, προσέχουμε τα θέματα της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, ότι γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές. Το θέμα της ποιότητας τώρα, προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι διάφορες πολιτικές έχουν ληφθεί υπόψη, ότι όλες οι απόψεις έχουν ληφθεί υπόψη και ότι δεν ε, ε, έχουμε τελευταία στιγμή ε, μια έκπληξη ότι κάτι έχει αφαιθεί κατά μέρος. Και υπάρχει και το θέμα του προγραμματισμού. Έχει να κάνει με το τι θέματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τι εξωτερικές δράσεις έχουμε αναλάβει, τι ισολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή Συναντήσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δυστυχώ όμω υπάρχουν περιπτώσει όπου έχουμε πολλέ διαρροέ εγγράφων. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στην ε, διαβούλευση εντό των υπηρεσιών. Και δεν πρέπει ένα πρωτοσχέδιο πρόταση να το θεωρήσει κανεί μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει ω είναι προϊόν συμφωνίας, ε, γιατί μπορεί να υπάρξουν εντωμεταξύ αλλαγές, ε, ε, ακόμα και από το σώμα των επιτρόπων. Οπότε όλο αυτό είναι τμήμα του κανονικού μου, του συνηθισμένου μου καθήκοντος και σας το λέω, γιατί με τους συναδέλφους μου πρέπει να εξασφαλίσω στην περίπτωση, ας πούμε, της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, ότι δεν έπρεπε να αρχίσει έρευνα πριν από την κατάλληλη στιγμή και ότι υπήρχαν κάποιες βέβαια ευαισθησίες οι οποίες ε, είναι ε, εύλογο να υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησαν όμως οι διαδικασίες και αυτή τη στιγμή υπάρχει πλέον ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η συγκεκριμένη πρόταση οδηγίας όσον αφορά τους κανόνες ε, έχουν γίνει σεβαστοί. Εμείς δουλέψαμε πάρα πολύ για να αποφασιστούν αυτοί οι κανόνες και δεν νομίζω ότι είναι λογικό να λέει κανείς ότι μόνο ε, το προτείνον τμήμα πρέπει να ακούσει τις διάφορες αντιπροσωπευτικές απόψεις. Η Επιτροπή έχει έναν πολύ ανοιχτό ε, τρόπο. Εμείς την ανάλυση μας τη δημοσιεύουμε, τις προθέσεις μας επίσης. παρουσιάζουμε χάρτες πορείας για τις μελέτες αντικτύπου, εξελόγησης αντικτύπου με σκοπό να προσελκύσουμε ε, τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, τους stakeholders. Θέλουν, θέλουμε να εισακουστούν οι απόψεις όλων. Αυτό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Δεν είναι ασυνήθιστο ο Γενικός Γραμματέας να ακούει πολλές ε, απόψεις πολλών εμπλεκομένων φορέων. Θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση να είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε τις απόψεις των ανθρώπων που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Το email που έστειλα τώρα σε Swedish Match 16 Οκτωβρίου ήταν απλώς μια ενημέρωση δημοσίως γνωστών ε, ε, πληροφοριών, γιατί είχε αρχίσει αυτό το θέμα ε, του Επιτρόπου Νταλή. Είχε γίνει στην αρχή μια ανακοίνωση προς τις Swedish Match και γι' αυτό θεωρούσα ότι έπρεπε να τους ενημερώσω ότι είχε ολοκληρωθεί η έρευνα και το email μου ήταν απλώς μια επιβεβαίωση αυτών που ήδη είχαν αναφερθεί στα ανακοινωθέντα τύπου. Δεν είπα τίποτε το καινούριο θεώρησα ότι έπρεπε να τους ε, πω ότι ε, ναι, επανέλαβα απλώς κάτι το οποίο ήταν ήδη γνωστό. Δεν ε, γνωρίζω τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του 2004 για τα καπνά, οπότε δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Γνωρίζω τη δουλειά του Αντιπροέδρου της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Εμείς προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες γενικές διευθύνσεις λειτουργούν σε επίπεδο ομάδων εμπειρογνωμόνων. Υπάρχει και σχετική έκθεση γι' αυτό. Είχαμε, είδαμε κάποιες πρακτικές που πρέπει κάπως να ενημερωθούν και να ευθυγραμμιστούν. Το δικό μου τμήμα συνεργάζεται με τον ε, αντιπρόεδρο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι, για παράδειγμα, ε, άνθρωποι που θεωρούνται ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες να είναι πράγματι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και να μην εκπροσωπούν μία ε, εταιρεία χωρίς αυτό να είναι γνωστό. Έχουμε λοιπόν μία διαδικασία. Όλες οι ομάδες εμπειρογνωμόνων εξετάζονται από αυτό το πρίσμα ώστε να σε, γίνονται σεβαστοί όλες, όλοι οι κανόνες της διαφάνειας. Τώρα η ομάδα υψηλού επίπεδου ε, με επικεφαλής του κύριο Στόιμπερ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά το 2014. Ε, θα υπάρξει μια νέα ε, ε επιτροπή το, στο τέλος του 2014. Μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να, να αποφασίσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Το γεγονός ότι σε μια ε, συνεδρίαση ο κύριος Στόιμπερ ε, υπέβαλε μια επιστολή ε, που είχε λάβει. Ε, αυτό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο, συμβαίνει ε, συχνά. Μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Συχνά συμβαίνει η ομάδα αυτή να λαμβάνει κάποια email κάποιες, για κάποιες ανεπίσημες απόψεις τις οποίες ε, ούτως ή άλλως θα δημοσιεύσουμε, στη συνέχεια στον ιστότοπο ε, της ε, ομάδας. Για να πω δηλαδή ότι δεν έγινε τίποτε το ασυνήθιστο και το γεγονός ότι αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι περίεργο, είναι τμήμα μιας κανονικής διαδικασίας των εργασιών της ομάδας. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ και στο ερώτημα το δικό σα, κύριε Πρόεδρε, για την αξιολόγηση αντικτύπου. Σα είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εξηγήσω και πάλι γιατί η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι στην καλύτερη θέση να προβαίνει σε αξιολόγηση αντικτύπου για τι ίδιε τι προτάσει τη. Πιστεύουμε ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λόγω του ότι άρχισαν να υπάρχουν οι μελέτε αξιολόγηση αντικτύπου και πιστεύουμε ότι η εξωτερική αξιολόγηση και από το ελεκτικό συνέδριο αλλά και από άλλους φορείς ε, έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η καλύτερη στον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Γιατί θεωρούμε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιολογήσουμε όλε μα εναλλακτικέ επιλογέ πριν φτάσουμε σε μία πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά θα σκότωνε το ίδιο το δικαίωμα πρωτοβουλία της, πρωτοβουλίας της εάν έδινε αυτό το, το, την αξιολόγηση αντικτύπου σε κάποιον τρίτο. Είναι τμήμα του τρόπου με τον οποίο αντισταθμίζουμε τα διάφορα ζητήματα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, σταθμίζει τα διάφορα κόστη και τα διάφορα ωφέλη μίας πρότασης και τελικά κάνει την επιλογή της για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξισορροπήσει αυτά τα, αυτές τις πτυχές. Αυτή τη στιγμή όμως έχει κάνει την επιλογή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπει ποιο συνδυασμό εναλλακτικών επιλογών θέλει να υποβάλει ως πρόταση, τότε βεβαίω είναι απολύτω δυνατό ε, εξωτερικοί φορείς να το εξετάσουν και να δουν κατά πόσο ε, συμφωνούν ε, ή θα ήθελαν μια διαφορετική επιλογή. Και Και ξέρουμε ότι υπάρχει και μία διεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ειδικά ασχολείται με την ποιότητα τη αξιολόγηση αντικτύπου και από την άλλη το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει από μόνο του κάποιες τέτοιου είδου αξιολογήσει, μελέτες που μπορεί να τις υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις χωρίς να κάνει η ίδια αυτή τη στάθμιση των ε, ε, διαφόρων συνεπειών γιατί πρέπει να έχει λάβει όλες αυτές τις πληροφορίες για να κάνει μια ενημερωμένη επιλογή, μια πολιτική επιλογή της ε, πρότασης που θέλει ή δεν θέλει να υποβάλει. Αυτή τη στιγμή γίνει λοιπόν η πρόταση και δημοσιευθεί όλοι μπορούν να δουν τα δεδομένα αυτά, τα οποία έχει συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά, στη συνέχεια, μπορούν ε, τρίτη φορείς ε, να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προβαίνει σε μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου. Τώρα, για το ερώτημα τώρα των πιστώσεων υποχρεώσεων. Ε, συμφωνούμε με τις ανησυχίες σας. Εμείς πάντοτε ζητούσαμε ένα ποσό για τις υποχρεώσεις αυτές σε ετήσια βάση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς που θα έρθουν. Είναι κοινή, ε, είναι, είναι ευρέως γνωστό ότι στο τέλος μιας ε, δημοσιονομικής περίοδου πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη αντιστοίχηση μεταξύ των ε, ετοιμάτων πληρωμών και των πραγματικών πληρωμών. Μα ανησυχεί το γεγονό ότι μπορεί να μην έχουμε αρκετά χρήματα να πληρώσουμε όλου του λογαριασμού. Έχουμε νομική υποχρέωση να ε, πληρώσουμε και έτσι αν. Αν δεν τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε, θα πληρώσουμε τόκους. Άμα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Παρά το γεγονό ότι έχουμε εξηγήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα στα κράτη-μέλη, συνεχώς μειώνουν τον αριθμό των ε, ε, πιστώσεων υποχρεώσεων για το προτινόμενο 5% περικοπές ε, στο προσωπικό. Ναι, έχουμε δει τι συνέπειε. γι' αυτό έχουμε προτείνει αύξηση του χρόνου εργασία από 37,5 σε 40 ε, ώρες την εβδομάδα για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε το, τη συνέπεια της μείωση του προσωπικού και κοιτάμε τι γίνεται και στου υπόλοιπα, υπόλοιπα όργανα για να μπορέσουμε συλλογικά να υπάρξει μια διαθεσμική αποτελεσματικότητα για να το πω έτσι, για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τον αντίκτυπο τη Νομίζω ότι τα απάντησα όλα. Αν ε, ξέχασα κάτι, ευχαρίστω να δευτερολογήσω, αλλά για την ώρα αυτά είχα να πω. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ντέι που απαντήσατε στις ε, ερωτήσεις και τώρα θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο, το συνάδελφο κύριο Πίπερ. Παρακαλώ κύριε Πίπερ, έχετε το λόγο. Κυρία Γενικέ Γραμματέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Ε, ορισμένοι συνάδελφοι μου ε, δημιούργησαν την εντύπωση μάλλον από τις ερωτήσεις που ετέθησαν αποκόμισε την εντύπωση ότι ε, σε ορισμένα απαντήσατε διεξοδικά αλλά όχι στη δική μου ερώτηση όσον αφορά την αξιολόγηση και τους δείκτες Είπατε ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις ε, για το θέμα αυτό με τα κράτη-μέλη, να δούμε τι θα γίνει με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτά τα θέματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντωμεταξύ βρίσκεται στη διαδικασία της ε, συναπόφασης. Και όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή πολιτική και στην γενικότερη αξιολόγηση, προφανώς και θα θέλαμε να ε, έχουμε και εμείς άποψη και θα το διεκδικήσουμε αυτό. Και κάτι άλλο. Έχει σχέση με το σε σύστημα, της μετακινήσεις. Και ρωτώ συγκεκριμένα, όταν λέτε ότι ναι μεν υπάρχει αυτός ο κανόνας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σε πόσες περιπτώσεις ε, έχει πράγματι προκύψει μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και πολύ συγκεκριμένη. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν ε, δεσμευτικά, νομικά δεσμευτικά κριτήρια που να επιβάλλουν τη μετακίνηση των υπαλλήλων. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, ο κύριος ε, Στάρς, ο Μπάρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε, αλλά σας είχα θέσει και κάποιες ερωτήσεις αφήσεις. Σας είχα ζητήσει να μου πείτε πέραν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστήλατε, εάν εσείς οι ίδια είχατε προσωπικές επαφές πέραν αυτού του mail. Επαφές είναι ένας όρος τον οποίο εσείς ορίζετε με τρόπο διαφορετικό, διότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον κύριο Περό φαίνεται πως δεν αποτελεί επαφή, αλλά εξαιρέσει αυτού του email. Έχετε επαφές με τη Swedish Match ή με κάποιους άλλους ε, του κλάδου και είχατε κάποια επαφή αναφορικά με τα παράπονα που είχαν εκφραστεί και αν ναι, τι ακριβώς συνέβη, τι υπόθηκε. Επίσης, το ηλεκτρονικό μήνυμα που στείλατε στον κύριο Περό αποτελούσε μια πρώτη, θα έλεγα, ενημερώσατε κάποιον για τα αποτελέσματα. Ήταν η πρώτη φορά που προβήκατε σε ένα τέτοιο διάβημα και κάτι ακόμα. Είπατε ότι κάποια στοιχεία δεν έτυχαν ε, ενδοϊπηρεσιακής συνεννόησης, διότι να ελέγχετε το ζήτημα της επικουρικότητας και δεν έγινε και εκ των υστέρων υπήρξε αυτή η ενδοϊπηρεσιακή διαβούλευση αλλά ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει ώστε από εδώ και στο εξή να μην υπάρχουν παρόμοιες διαρροές διότι αν φοβούμεθα διαρροές τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπου θα καθυστερούν και άλλα νομοθετικά κείμενα. Κυρία Κρέσλε, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις δίκιο έχετε. Ε, στη σελίδα 40, στην ερώτηση 44 μου ξέφυγε το θέμα των παραρτημάτων. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της ε, κινητικότητας. Ποιοι γενικοί διευθυντές παρέμειναν στη θέση τους πάνω από 7 χρόνια. Το επόμενο ερώτημά μου αφορά αυτό που είπε και ο κύριος Στάρς, δηλαδή τις δικές σας τις ε, πρωτοβουλίες σχετικά με την οδηγία για τον καπνό. έχουμε εκείνους ε, οι οποίοι επεξεργάστηκαν την Συμφωνία για τον Καπνό το 2004 και λένε βεβαίως ότι ως προϋπόθεση ήταν ανέκαθεν σαφές ότι ίσχυε ότι δεν θα αλλάξει αυτή η οδηγία του καπνού. Αυτό είναι και μια προϋπόθεση που είχε θέσει η βιομηχανία καπνού και το καταλαβαίνω, δεν θα κάνει κανείς μια τεράστια επένδυση χωρίς να ξέρει αν θα παραμείνει ενισχύ νομική βάση. Και η δική παρέμβαση πάντα με εντυπωσίαζε γιατί έλαβε χώρα όταν έτρεχαν ήδη οι ανακρίσεις για τον κύριο Νταλή. Θεωρώ ότι είστε έξυπνοι υπάλληλος. και όταν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση ε, κανονικά δεν κάνει κανείς τίποτα εκτός αν εξαναγκαστεί. Γι' αυτό λοιπόν για μένα αυτή σας η παρέμβαση είναι ακατανόητη και δεν την καταλαβαίνω. Εκτός εάν θυμηθεί κανεί ότι αυτό η σταθερότητα στην ε, νομοθεσία αποτέλεσε κατ' ουσία και τη βάση της όλης υπόθεσης. Μετά, το θέμα με τα λόμπι. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ε, οι ε, σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εταιρείες ε, καπνού. Ρώτησα ποιος πέρασε από την Κομισιόν σε ομάδες πίεσης και αντίστροφα. Δεν μου απαντήσατε. Εγώ όμως σας είπα τουλάχιστον πέντε ονόματα υπαλλήλων που πέρασαν στη βιομηχανία καπνού. Και ρωτώ, τους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τις ομάδες πίεσης τους βρίσκεται επαρκής εμείς ε, έχουμε θέσει κάποιες προϋποθέσεις ε, που ακόμα όμως δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. Αυτούς λοιπόν τους κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή τους θεωρείτε ε, ικανοποιητικούς ή όχι. Κατόπιν, πώς θα πρέπει να επιτύχουμε αυστηρότερες Τυπικέ διαδικασίες. Ε, στις δημόσιες συμβάσεις, εκεί υπάρχουν πάρα πολλέ σχέσει με τις ομάδες επίσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε οι υπάλληλοι να αλλάξουν τους κανόνες. Εσείς το σκέφτεστε αυτό. Και πάω στο ερώτημα υπαριθμών 36, δηλαδή στο ερώτημα των συναντέλφων κατά πόσον είσαστε ενημερωμένοι για την εξέλιξη των ανακρίσεων στην περίπτωση Νταλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμεί, λέει ο πρόεδρο, Και τελευταίο ε, ερωτών ο κ. Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Στις απαντήσεις σας διαβάσαμε ότι το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων δεν είναι επίκαιρο, δεν εφαρμόζεται κλπ. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα αποτελέσματα, μόνο τα διδάγματα τα οποία συνάγονται μετά από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και αν η σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι πλέον επίκαιρο ζήτημα, τι γίνεται, ότι δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να προκύψουν παρόμοια προβλήματα, η Κομισιόν είναι ερμητικά κλειστή σε παρόμοιου είδους δραστηριότητες. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα συμπεράσματα και τα διδάγματα που συναγάγατε. Ευχαριστώ. vielen Dank. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο ε, τον λόγο. Ε, κατόπιν τούτου, κυρία Γενική Γραμματεία, θα ήθελα να σα δώσω το λόγο για να απαντήσετε εσεί τι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Φυσικά γνωρίζω τον ρόλο του Κοινοβουλίου, γι' αυτό λοιπόν αναφέρθηκα στην ε, ε, διαθεσμική συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει πριν να κρίνουμε την επιδόσεις. Συμφωνώ απόλυτα και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν υπενθυμίζει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο καθημερινά. Το Κοινοβούλιο έχει τα ίδια δικαιώματα για να ορίσει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ζήτημα είναι ότι η Κομισιόν χρειάζεται το πλαίσιο πρώτα να συμφωνηθεί, πρώτου να ε, προχωρήσουμε στην παρακολούθηση. Να κάναμε ό,τι ήταν στις δυνατότητές μας για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου και τώρα τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις και μόλις αυτές οι αποφάσεις ληφθούν τότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το έργο μας. Και όπως υπόθηκε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη, όπως είπε και το Ελεκτικό συνέδριο. Και δεν πρέπει να παραμιλήσουμε την ανάγκη διασφάλισης νομιμότητας και ε, τυπικότητας. Θα ήθελα να κάνω έκκληση προς το Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει με το πλαίσιο και να μπορέσουμε να έχουμε ένα όσο πιο απλό πλαίσιο για να είναι πιο εύκολο να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Ακούσαμε τα παράπονα τα οποία προβλούνται από ενδιαφερόμενους ότι είναι πολύ δύσκολο να συμμορφωθούν, δίνει χώρο σε παρανοήσεις, θα πρέπει λοιπόν να απλουστευτεί. Γι' αυτό και έκανα έκκληση για μια διαθεσμική συνεργασία. Δεν έχω ενώπιον μου, διότι δεν είμαι ο γενικός διευθυντής για τους, ανθρώπινου ανθρώπινους πόρους. Δεν ξέρω τι, ε, τι αλλαγές έχουν γίνει στο ε, θέμα της κινητικότητας. Ε, παρά λέω ότι ο γενικός κανόνας είναι η κινητικότητα και αυτό λαμβάνει υπόψη όταν απαντάω στις ερωτήσεις, είναι ο γενικός κανόνας, εντάξει μπορούν να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις και είναι οι επίτροποι οι οποίοι αποφασίζουν πώς θα διορίσουν τους γενικούς γραμματές και πότε θα πρέπει να τους ε, να εφαρμόσουν σε αυτούς τους γενικούς διευθυντές την κινητικότητα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν, δεν είχα προ... επαφές με τους εκπροσώπους του βιομηχανής καπνού. Η μόνη επαφή που είχα με τη Swedish Match ε, αφορούσε ισχυρισμούς που έκαναν για τον Πίτρο Πονταλή και η μοναδική επαφή μου ήταν όπου τους είπα ότι ε, έστειλα την υπόθεση στην Όλαφ ε, και οι επαφές που είχαν οι υπηρεσίες μου έχουν ήδη ε, μπει στα πρακτικά και υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα πως θα να γνωρίζω πως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την διαρροή κάποιων εγγράφων είναι κάτι, ένα πρόβλημα το, της σύγχρονης εποχής, όπως γνωρίζετε. Αν υπάρχουν καλές ιδέες, πώς, καλές ιδέες για το πώς θα αποφεύγουμε αυτές τις διαρροές, παρακαλώ είμαι στη διάθεσή σας και θα ήθελα να τις ακούσω. Οι Επίτροποι έχουν γνωρίζετε την δυνατότητα να συζητούν μαζί μεταξύ τους διάφορα πράγματα, τα οποία όμως δεν βλέπουν ποτέ το φως δημοσιότητας, ε, αλλά γράφονται σε ένα χαρτί, ε, διαρρέει το χαρτί και βγαίνει ως ε, πρόταση της Κομισιόν για το χύψη ε, θέμα, ενώ η ίδια Κομισιόν δεν προτίθεται να ε, προβεί σε μια τέτοια ανακοίνωση. Όπως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο με τον ε, μέσα τα οποία διαθέτουμε σήμερα να γνωρίζουμε πού προέρχονται οι διάφορες διαρροές. Δεν μπορώ να πω για τη συμφωνία περί καπνού 2004, δεν ε, συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις, άρα δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω. Τώρα. Στην Κομισιόν υπάρχουν κανόνες σχετικά με την ε, με τις εργασίες ε, των ε, υπαλλήλων, με τα καθήκοντά τους κλπ ε, και τα πρόσωπα τα οποία εγκαταλείπουν την Κομισιόν θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν άλλες εργασίες, δεν θα πρέπει η Κομισιόν να παρεμποδίσει περαιτέρω εξέλιξή τους εκτός της Κομισιόν και αυτό εφαρμόζεται. Οι κανόνες λοιπόν είναι αυστηροί και εφαρμόζονται. Λυπάμαι που δεν απάντησα στην ερώτηση σχετικά με τις ε, υπηρεσίες, ε, με τις agents. Έχουμε καταλήξει μια συμφωνία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Ε, λάβουμε υπόψη τις συστάσεις ε, του ελεκτικού συνεδρίου για το ζήτημα των ε, υπηρεσιών, ε, των agencies, αλλά η Κομισιόν δεν είναι υπεύθυνη για αυτές τις υπηρεσίες και αυτό που κάναμε είναι να εφαρμόσουμε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια κοινή προσέγγιση και πρέπει να εξετάσουμε κάποιες περιπτώσεις όπου τα διοικητικά συμβούλια ορίζουν κάποιους επιστήμονες φορτίζουμε ναι, φροντίζουμε και στην περίπτωση αυτή να μην προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων και η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις ε, αναφορικά με ε, θέματα αυτές της συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια αυτών των υπηρεσιών με βάση τη συμφωνία που έχουν συνέβη με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ja, vielen äh, Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν συμπληρωματικέ ερωτήσει, κυρία Γκρέσλερ. Ναι, επανέρχομαι στην ερώτηση αριθμού 44. Διότι εδώ ρωτάμε πόσοι υπάλληλοι δεν συμμετείχαν σε κάποιο διαγωνισμό. Γιατί δεν απαντήσατε στο ερώτημα, διότι στο παράρτημα εδώ δεν γίνεται διάκριση όλων των βαθμών, όλων των βαθμίδων των συμμετεχόντων. Και αυτό το οποίο κρύβεται πίσω από την ερώτηση είναι διότι συχνά εδώ πρόκειται για υψηλόβαθμους αξιωματούχου οι οποίοι προσλήφθηκαν εκτός διαγωνισμού. Και θα ήθελα να σα ε, ξαναζητήσω να απαντήσετε στο ερώτημά μου και σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ε, ο, ο συνάδελφος ε, θέλει να πει κάτι. Ναι, διαπίστωσα πως μια ερώτηση που έχει από την κυρία Βρέσλερ σχετικά με τον κύριο Πετίν. Νομίζω ότι δεν λάβαμε απάντηση σε αυτό το θέμα. Ο Πρόεδρος, ναι, ευχαριστώ. Άλλος επιθυμεί να παρέμβει. Όχι. Κανένα μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θέλει να θέσει ερώτηση, να θέσω εγώ που έχει άμεση σχέση με, με ευθύνη του κυρίου Λιμπεράτσκι για την προστασία ε, κατά τη διαφθορά σου. Δεν ε, μάλλον γνωρίζετε ότι έγινε η παρέτηση του κυρίου Νταλή και στην Επιτροπή μας εξετάσαμε τις συνθήκε κάτω από τις οποίες παρετήθηκε αλλά και τις συνέπειες, τα διδάγματα που πρέπει να συνάγουμε από αυτήν την κατάσταση. Ένα κοινοβούλιο εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία και θα πρέπει να ελέγχει την δίκηση. Πρέπει να θέτει ερωτήσεις, να απαιτεί εξηγήσεις. Ο πρόεδρος Σούλτ έθεσε στον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόζο, τα σχετικά ερωτήματα. Θα δούμε ποιες θα είναι οι προφορίες που θα λάβουμε, οι απαντήσεις θα δοθούν στους άμεσα εκλεγμένους βουλευτές τώρα σε ό,τι φορά τον κώδικα δεοντολογίας και τον αγώνα κατά της ε, διαφθοράς θέλαμε την προσωπική σας άποψη. Έχετε την ε, εντύπωση ότι το όλο σύστημα, υπάρχουν σύστημα είναι επαρκές για να ελέγχονται οι επίτροποι αλλά και όλοι οι συνεργάτες της Κομισιόν και παράλληλα πώς μπορούν να προστατεύονται από τις ε, επιρροές που μπορούν να τους ασκούνται από το εξωτερικό. Στη Γερμανία τα, συνεργάτες να είχαν προστασίες από, την, από εξωτερικές επιρροές. Θα μπορούσατε λοιπόν κυρία Ντέι να μας ε, πείτε για τον επαρκή ή ανεπαρκή χαρακτήρα των κανόνων που ισχύουν και σε ό,τι φορά τον, ε, το πλωστάσιο που υπάρχει δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από μέλη. Σας καλώ κυρία Ντέι να απαντήσετε σε ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Well, starting... Ευχαριστώ. Θα αρχίσω από την τελευταία ερώτηση. Πιστεύω ότι ο κώδικας διοντολογίας που ισχύει για τους επιτρόπους είναι πάρα πολύ αυστηρός και Πιστεύω ότι αν δει κανεί ε, τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη, και υπάρχουν και διαφορέ αν δει κανεί τι ισχύει σε διάφορου διεθνεί οργανισμού και στα άλλα κράτη-μέλη, νομίζω ότι ο ε, κώδικα διοντολογία Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μάλλον αυστηρό και πρέπει να σα επιβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ αυστηροί ένας από τους κύριους τομείς ε, για τους οποίους ισχύει είναι σε περίπτωση επιτρόπων που έχουν φύγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μια περίοδο μάλιστα δεν μπορούν να αναλάβουν άλλα καθήκοντα σε άλλο επάγγελμα αν δεν έχουν υποβάλει ε, την ε, υποψηφιότητά τους ε, για αυτό το νέο επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει ε, στους επιτρόπους και όχι σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους ε, άλλων κοινοτικών οργάνων. Οπότε πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέπεται από τον αυστηρότερο κώδικα δεοντολογίας και από τους αυστηρότερους κανόνες. Για το ερώτημα τώρα του ρόλου του Μισελ Πετή, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Ο κύριος Πετή έφυγε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007, ε, σεβόμενος πλήρως τους κανόνες για τους πρώην ε, ε, υπαλλήλου. στο γεγονός ότι το 2012 δουλεύει κάπου αλλού, νομίζω ότι είναι κάτι το πάρα πολύ λογικό για κάποιον που έφυγε πριν από την Επιτροπή πριν από πέντε χρόνια. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι περαιτέρω πληροφορίες θέλετε από μένα, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουμε τους κανόνες. Έχουμε απαντήσει και γραπτός και προφορικός σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη θέση του ε, μετά από την ε, θητεία του στην Επιτροπή. Ευχαρίστω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας, κυρία Γκρέσλε. 44 ερώτηση λέτε πόσε θέσει ε, έχουν καλυφθεί από επιτυχημένου από επιτυχημένους ε, διαγωνιζόμενους ε, σε διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας έχω απαντήσει. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, ευχαρίστως να τις ε, υποβάλουμε και αυτές. Αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου τα δεδομένα αυτά που ζητάτε. Αν λείπει κάτι, ευχαρίστως να σας το διαβιβάσω κάποια στιγμή σε μεταγενέστερο στάδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι μας είπατε θα μας απαντήσετε γραπτά και κατόπιν τούτου προτείνω ε, σε γραπτή μορφή να διευκρινίσουμε και εμείς τις ερωτήσεις μας και να σας τις διαβιβάσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ζητήσει άλλοι ε, τον λόγο και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή κατά πόσον θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου. Μήπως υπάρχει κάποιος ε, να θέλει να λάβει το λόγο. Από ό,τι φαίνεται όχι. Κατόπιν τούτου σας ευχαριστώ θερμά κυρία Γενική Γραμματέα για την επίσκεψή σας εδώ και επίσης ε, και για την τοποθέτησή σας ε, στα ερωτήματά μας. Και τα λέμε. Γεια. Κλείνει λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσια διάταξης, το 12 και πάμε στο επόμενο θέμα, το 13. Πρόκειται για ειδική έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνεχής για τη συγχρηματοδότηση. Η συγητής είναι ο κύριος Μπόκουσλαφ Λιμπεράτσκι και εκ μέρου ε, του ελεγκτικού συνεδρίου να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Οβίδιο Ισπύρ. Και θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω τον εισηγητή κατά πόσον θέλει να λάβει το λόγο εισαγωγικά ή να μιλήσει καλύτερα το ε, πρώτα το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία αυτής της έκθεσης. Πρόκειται για μια έκθεση ιδιαίτερα σημαντική, όπου παρατηρούμε να υπάρχει ένας ε, σημαντικός, μεγάλος επαγγελματισμός ε, για την επαγγελματικότητα. Πρόκειται για, τα, για τους λιμένες και τονίζουμε επίσης την αποτελεσματικότητα. Αυτό το οποίο ε, συμβαίνει εδώ είναι ότι αναφέρονται και τα θετικά παραδείγματα αλλά και τα αρνητικά. Υπάρχουν λίγα θετικά παραδείγματα και γι' αυτό θα πρέπει να τα προωθήσουμε και να τα προβάλλουμε. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα ε, παραδείγματα τα οποία χρειάζεται να αποφύγουμε. 27 ε, προγράμματα εξετάστηκαν, 7 δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά. 4 χώροι εξετάστηκαν που λαμβάνουν 85% των πόρων για προγράμματα που αφορούν του θαλάσσιου λιμένες ε, για την περίοδο 2000-2006. Ευχαριστώ που επιλέξατε αυτήν την, αυτόν τον προσανατολισμό για την ανάλυση. Υπάρχουν κατηγορίες ε, για τις οποίες ε, υπάρχουν ε, ελλείψεις, υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα προγράμματα τα οποία δεν έχουν προοπτική η έκθεση του Ελληνικού Συναδρίου έχει, είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση της Κομισιόν. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Αυτή η ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου μας έδειξε ότι η Κομισιόν έπρεπε να οργανώσει την παρακολούθηση της δαπάνης των ταμείων. Από πλευράς Κομισιόν υπήρξε κάποια παθητικότητα θα έλεγα, αλλά τώρα πια έχει προλάβει και αντιδράσει. Θα σχολιάσετε αυτό το σημείο και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς το ελεκτικό συνέδριο. Σε ένα περίπου χρόνο θα έχουμε φτάσει στο τέλος ε, των ε, δημοσιονομικών ε, προβλέψεων και θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Να... Διότι αν λάβουμε έκθεση για την προηγούμενη περίοδο, την εξετάζουμε την τελευταία χρονιά των που αφορούν τις διαφορές δημοσιονομικές προβλέψεις και έτσι καθυστερούμε. Ευχαριστώ κύριε Λιμπεράτσκι. Το ελεκτικό συνέδριο έχει το λόγο. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, dear chairman, dear honorable members. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Χαίρομαι όλου ιδιαίτερω που βρίσκομαι εδώ σήμερα να συμμετέχω στη συζήτησή σα για το σχέδιο εκθέσεω που έχει ω θέμα την ειδική έκθεση υπαριθμών 4 του 2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρήση διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχή για τη συγχρηματοδότηση υποδομών μεταφορών στι θαλάσσιους λιμένες» είναι μια αποτελεσματική επένδυση. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που, βρίσκω, που βλέπω ότι ε, καλωσορίζει ο κύριος Λιμπεράτσκι, ο εισηγητής, ε, την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις επενδύσεις θαλάσσιους σημαίνες μέσω των ταμείων των διαρθρωτικών, των ταμείων συνοχής. Είναι σημαντικό αυτό στο πλαίσιο της περίοδου 2000 με 2006 που ήταν ο στόχος του ελέγχου μου, 2,8 ε, εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία αυτά διατέθησαν ε, σε, ε, στις υποδομές αυτές. Επιπλέον 3,4 δις ευρώ προχρηματοδοτήθηκαν για την περίοδο 2007 έως 2014. Σκοπό είχαμε να δούμε πόσο αποτελεσματικές ήταν αυτές οι, αυτές οι υποδομές, πόσο αποτελεσματική ήταν αυτή η επένδυση ε, κατά πόσο δηλαδή ολοκληρώθηκαν οι στόχοι και ε, ήταν σωστά τα αποτελέσματα. Επικεντρωθήκαμε σε 27 προγράμματα στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Χώρες που λαμβάνουν πάνω από 85,5% των ε, χρημάτων για τους θαλάσσιους λιμένες κατά την προγραμματική περίοδο. Θα σας πω τι διαπιστώσαμε. Καταρχάς, ε, αναρωτηθήκαμε κατά πόσο τα προγράμματα είχαν τους κατάλληλους στόχους ε, και, αν είχαν επειδή είχαν επιλεγεί για χρηματοδότηση από τον προπολογισμό, ε, ελπίζαμε να υποστηρίζουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους πολιτικής μεταφορών. Όμως μόνο τα δύο τρίτα πληρούσαν αυτό το κριτήριο. Επτά είχαν άλλους στόχους και δύο είχαν στόχους στόχους που θεωρούσαν ότι ε, θεωρήσαμε εμείς ε, στο ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν ήταν ε, η κατάλληλη και συμβατή. Ήταν μεικτά τα αποτελέσματα. Σε σχέση με το έγκυρο, 41% των προγραμμάτων ολοκληρώθηκαν εγκαίρως, αλλά 44% των προγραμμάτων παρουσίασαν καθυστερήσεις, με μέσο όρο καθυστέρησης τους 26 μήνες τέσσερις από, ε, τέσσερα από τα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή του ελέγχου. Το προφανές επόμενο βήμα ήταν να, δει, να δούμε τι χρήση έγινε των 23 ε, προγραμμάτων που είχαν ε, ολοκληρωθεί. Μέχρι τα μέσα του 2010, όταν έγινε ο έλεγχος, 19 χρησιμοποιούνταν. Τρία δεν χρησιμοποιούνταν και ένα είχε μόνο λειτουργούσε μόνο εν μέρη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των υποδομών αυτών. Ε, οι ελεγκτές ήταν τη απόψεω ότι χρειάζονταν περισσότερη επένδυση πριν ε, να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως αποτελεσματικά. Από τα 23 ολοκληρωμένα προγράμματα, τα 11 υποστήριζαν τους σωστού στόχου των μεταφορών, 4 ήταν εντελώ αναποτελεσματικά και 3 ε, τρία δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου. Ήταν ανεπιτυχής, ε, δηλαδή τα προγράμματα. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις, ε, δεν είχαν ολοκληρωθεί ε, οι κατασκευές, κάτι το οποίο ε, ήταν ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε σχέση με το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των θαλασσίων. Δεν είχαν γίνει, των θαλασσίων λιμένων, δεν είχαν γίνει οι κατάλληλες αξιολογήσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Λιμπεράτσκι έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη προγραμματισμού των αναγκών αναγκών πριν γίνουν τέτοια έργα. Σε σχέση τώρα με τη διαχείριση, είχε δοθεί λίγη προσοχή στην παρακολούθηση και την εποπτεία των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, με επιτροπέ παρακολούθηση και διαχειριστικέ αρχέ να εστιάζονται στο ποσοστό των δαπανών ε, αντί για τη χρήση και την αποτελεσματικότητα. Οι δείκτε σκοπό είχαν να παρακολουθήσουν μόνο την απορρόφηση και το επίπεδο των κατασκευών, αλλά υπήρχαν λίγα αποδεικτικά στοιχεία ότι Ευρωπαϊκή, ότι η Επιτροπή ε, παρενέβει στις επιτροπές παρακολούθησης για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική ε, χρήση των κονδυλίων για τα επτά μεγάλα προγράμματα ε, και τα προγράμματα που ε, πήραν χρηματοδότηση από τα ε, Ταμεία Συνοχής. Θέλουμε λοιπόν να προβούμε σε κάποιες συστάσεις, να υπενθυμίζει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη την υποχρέωσή τους να χρησιμοποιούν τα κονδύλια με τρόπο συμβατό με την οικονομική διαχείριση, Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι όροι σε σχέση με την στρατηγική, την μακροπρόθεση τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη λιμένων. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τη χρήση ε, των δικτών ε, αποτελεσμάτων και αντικτύπου από τι διαχειριστικέ αρχέ και να ενισχύσει τι διαδικασίε αξιολόγηση για να βελτιώσει την ανείχνευση σοβαρών αδυναμιών και επίση ε, την ανάληψη διορθωτική δράση. Με ενθαρρύνει το γεγονό ότι ο εισηγητή υποστηρίζει τι συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου και ε, προτείνει ακόμη περισσότερες συστάσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ε, προβλήματα με την ε, κακή χρήση των κονδυλίων στο μέλλον. Χαίρομαι που συμφωνεί ότι πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι και ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση ε, των αποτελεσμάτων και ε, των συνεπειών που είχαν οι κατασκευές των υποδομών αυτών. Η παριθμόν 4 έκθεση του 2012 έλαβε θετικά σχόλια από τη δημοσίευσή της, επικροτήθηκε ιδιαίτερα. Ε, ελπίζουμε να ακούσουμε επικοδομητικές συστάσεις. Πρόκειται για συστάσεις τις οποίες είδαμε στη δουλειά του εισηγητή και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε έτσι να συμμετέχουμε σε καλύτερη οικονομική διαχείριση των κατασκευών αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ το ελεκτικό συνέδριο, λέει ο Πρόεδρος, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στην κυρία Μαρεάτη από τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειών. Έχετε το λόγο. Στον κύριο Μαριάτη, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ε, να πω ότι η Κομισιόν ε, διάβασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ε, έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και ευχαριστώ τον κύριο Σπύρ για την παρουσίασή του εδώ. Η επεξεργασία αυτής της έκθεσης είχε ως αποτέλεσμα σε, την σεβάθουσα ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, οι οποίες συνεχίζουν να εφίστανται. Πάντως η έκθεση αυτή αποτελεί μια διάγνωση της κατάστασης και επιτρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Οι απαντήσεις που έδωσε η Κομισιόν ε, μας έκανε να διαπιστώσουμε ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη μπει στα σκαριά και η Κομισιόν μετά από την έκθεση αυτή επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για να ε, λάβει υπόψη τη τις συστάσεις του συνεδρίου και την οργάνωση επισκέψεων. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λιμπεράτσκι για την έκθεση που συνέταξε και αυτό σημαίνει το Κοινοβούλιο να πάνε υπόψη όλες τις δράσεις που έχει αναλάβει η Κομισιόν για την αποτελεσματικότητα των δράσεων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτού να περάσω στι συστάσεις αυτέ καθεαυτές με δύο παρατηρήσει προκαταρκτικού χαρακτήρα. Η πρώτη αφορά σε θέματα χρονοδιαγράμματος. Οι αναλύσεις που έγιναν αντικείμενο της έκθεσης ε, του συνεδρίου ε, καταρτήθηκαν το 2009 και τώρα βρισκόμαστε το 2013. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν τα προγράμματα θα πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω Αφετέρου, τα σχέδια τα οποία μελετήθηκαν ε, αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2000-2006, δηλαδή την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αφορούν εκείνη την περίοδο. Η περίοδο του 2007-2013 περιλαμβάνει μια σειρά βελτιώσεων, ειδικά για την έγκριση κάποιων προγραμμάτων από την Κομισιόν. Για την επόμενη περίοδο 2014-2020, η Κομισιόν πρότεινε κάποιες βελτιώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και για τις οποίες μίλησε ο κύριος Ισπύρ. Η δεύτερη παρατήρηση είναι εξή. Οι παρατηρήσεις που αποτελούν αντικείμενο του συνεδρίου είναι ε, αφορούν κοινέ δράσει και έτσι ο έλεγχο εμπίπτει στην ευθύνη των κρατομέλων. Η Κομισιόν δεν πρέπει να αποφασίζει η ίδια παρά μόνο σε ό,τι αφορά τα μεγάλα προγράμματα, δηλαδή προγράμματα που έχουν ένα κόστο υψηλότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επί των 27 προγραμμάτων μελέτησε το συνέδριο, μόνο 7 εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή μεγάλα προγράμματα άνω των 50 εκατομμυρίων. Τα... Εδώ μιλάμε για δεκάδες ε, εκατοντάδες προγράμματα. Δεν μπορούν λοιπόν ως αυτού να παρακολουθηθούν από τις ε, επικομισιόν αλλά από τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες των ε, κρατομελών και διαχείρισης και γίνονται συχνά και τακτικά επισκέψεις και έλεγχοι. Η Κομισιόν θα ήθελα να τονίσω ότι στα 27 από τα προγράμματα που ελέγχθηκαν, 19 είχαν ολοκληρωθεί και ήταν λειτουργικά όταν έγινε η επίσκεψη του συνεδρίου. Το, αυτό σημαίνει ότι το 70% των προγραμμάτων ήταν αποτελεσματικά. Αν κάνουμε σήμερα την ανάλυση, ε, τέσσερα από τα προγράμματα τα οποία ήταν ατελή όταν έγινε η επίσκεψη του συνεδρίου, από αυτά απομένει μόνο ένα σχέδιο που δεν έχει ολοκληρωθεί. Να υπενθυμίζω ότι οι καλύτερε γραμμέ για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 2000-2006 προβλέπει πω τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα προγράμματα μέχρι το Σεπτέμβριο 2012 που ήταν η ημερομηνία η οποία είχε οριστεί στις κατηδίες γραμμές που ενέκρινε η Κομισιόν για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 2006 για τις συστάσεις τώρα του κ. Λιμπεράτσκι και να, θα ήθελα να δηλώσω ότι η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα με το ότι χρειάζεται καλύτερη ε, δημοσιονομική διαχείριση ε, της παρέμβαση ιδιαίτερα στον ε, θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Τώρα η πρώτη σύσταση και η δεύτερη που συνδέονται σε ό,τι αφορά τους δείκτες ε, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. Να πω ότι για περίοδο 2006-2013 μεγάλα προγράμματα που ενέκρινε η Κομισιόν περιλαμβάνουν ήδη δείκτες υλοποίησης και αποτελεσμάτων. Αυτοί οι δείκτες έχουν καθοριστεί σε επίπεδο προγραμμάτους και ξέρετε ότι σε περίπτωση κοινή διαχείρισης αυτοί οι δείκτες καθορίζονται σε επίπεδο προγραμμάτων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του βασικού άξονε των προγραμμάτων αυτών. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων, μια παρατήρηση λογική. Δηλαδή, για να κάνουμε αξιολογήσει χρειάζεται να παρέλθει κάποιο χρόνο για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Κάναμε μια αξιολόγηση για την περίοδο 2014-2019 που έγινε το 2012. Χρειάστηκε να περιμένουμε πέντε χρόνια για να μπορέσουμε λοιπόν, να έχουμε τα, τη δυνατότητα να προβούμε στην εξέταση αυτών των προγραμμάτων. Τρίτη σύσταση που αφορά τη μέση διάρκεια και την ποιότητα των διοικητικών διαδικασιών. Η Κομισιόν τονίζει πως ε, μαζί με τις Εθνικές Αρχές Διαχείρισης έχει δημιουργήσει διάφορα εργαλεία για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα διοικητικών διαδικασιών. τέταρτη σύσταση προτείνει να αποκριστεί η πληρωμή όταν ε, ε, υπάρχει κακοδιαχείριση, είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε. Πέμπτη σύσταση προτείνει να βελτιωθεί η ενημέρωση σχέση με την πρόοδο των εργασιών. Εδώ η Κομισιόν θα συνεχίσει να εξετάζει τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή τη για την περίπτωση κοινή διαχείριση. Θα μπορεί να το κάνει στο πλαίσιο διμερών και τεχνικών ε, συναντήσεων και επαφών και όλες τις δυνατές επαφές ε, επί τοπίως. Σε όλη την έκτη, την έκτη σύσταση, προτελευταία δηλαδή, που προτείνει ανάλυση του προσανατολισμού και ε, ευαισθητοποίηση των κρατών μελών σε θέματα ε, δημοσιονομική διαχείριση, να πω ότι η Επιτροπή Ρέτζο έχει αποκτήσει νέα εργαλεία για να βοηθήσει τις ε, εθνικές αρχές και η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη αυτήν την παρατήρηση και θα επαληθεύσει την δυνατότητα εφαρμογή στην πράξη αυτή τη ανάλυση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτών των νέων λουτιωριών. Και τελευταία σύσταση που προτείνει να τροποποιηθούν ε, κανονισμοί για να μπορέσει η Κομισιόν να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο στι επιτροπέ παρακολούθηση. Η Κομισιόν ε, συμμερίζεται αυτή την άποψη για την ενίσχυση του ρόλου της στις Επιτροπές Παρακολούθησης, αλλά τονίζει ότι ο ρόλο της Κομισιόν δεν περιορίζεται μόνο στις επιτροπές παρακολούθησης αλλά ε, και σε άλλα, από άλλες συναντήσεις προβλέπω του κανονισμούς, ετήσιε συναντήσεις, διμερείς με τι εθνικές αρχές και περιφερειακές αλλά και μια μόνιμη επαφή με τις επιτροπές διαχείριση που επιτρέπει να προοδεύσουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν στο πλαίσιο του νέου ε, κανονιστικού πλαισίου η Κομισιόν προτείνει νέα μέσα για την καλύτερη εφαρμογή αυτής της πολιτικής, την μεγαλύτερη επικέντρωση στους στόχους, ένα πλαίσιο πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό κλπ. Για να ολοκληρώσω, να πω ότι παραμένουμε στην διάθεσή σας ε, για να απαντήσω σε δεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ε, πρώτος ε, είχε ζητήσει το λόγο ο κύριος Σκυλακάκης, ο οποίος όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Έχουμε λοιπόν την κυρία Ότης και μετά τον συνάδελφο κύριο Σταυρακάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τα μέλη του Λευκού Συνεδρίου και της ε, Κομισιόν. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο για αυτήν την ειδική έκθεση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των διαστοντικών πόρων και της συνοχής ε, στην χρηματοδότηση ε, έργων για τους θαλάσσιους λιμένες και συμφωνώ με την έκθεση Λιμπεράσκη. Συμφωνώ επίση με το σύνολο των συστάσεων ε, που γίνονται τόσο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και προ τα κράτη-μέλη, που είναι και η βασικοί της, ε, για την υλοποίηση των προγραμμάτων και για την καλή διαχείριση των ε, ποσών που έχουν επενδυθεί. Τα λιμάνια θεωρούνται ότι παίζουν μεγάλη ρόλο για, στις εθνικές οικονομίες και απαιτούν μεγάλες επενδύσεις. Θα ήθελα να ε, ζητήσω, να δηλώσω ότι υπάρχει ανάγκη αυστηρών ελέγχων. Πέραν τούτων, από ε, την Κομισιόν ακούσαμε τις διαφορετικές δημοσιονομικές περιόδους ε, εξετάζουμε το 2006 βρισκόμαστε το 2013. Ευτυχώς ε, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για το θέμα υλοποίηση ε, υλοποίησης ελέγχων πιο αποτελεσματικών που οφείλονται και στο πρόγραμμα δράσης Κομισιόν του 2008. Είναι λοιπόν θετικό το να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι ελλείψεις που υπήρχαν βελτιώνονται και πως ε, θα πρέπει να δώσουμε πολύ βάση σε αυτές, τους ελέγχους. Τώρα, η Επιτροπή και οι ελεγχτικές ελληνικές αρχές θα πρέπει να ασκούν πλήρως ε, το έργο τους. Μία από τις ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πως ε, όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν, εάν υπάρχουν κάποια τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και υπάρχει αδυναμία ολοκλήρωσης κάποιον εξ αυτών. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο, ο συνάδελφο κ. Σταυρακάκη. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ καλό σχέδιο έκθεση που έχει υποβάλει, καθώ ο ίδιο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο και ενήμερο σε θέματα σχετικά με τι μεταφορέ. Αναμφίβολα οι παρατηρήσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου στη συγκεκριμένη έκθεσή του οφείλουν να μα προβληματίσουν, εφόσον συμπεραίνουν ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχή για έργα υποδομή μεταφορών στα θαλάσσιους λιμένες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που παραθέτει το Ελεκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του, για το οποίο η Επιτροπή έχει εγείρει αντιρρήσει. Αναφέρομαι στην υπόθεση κατασκευή Μαρίνα στη Μητυλίνη, ένα από τα ελληνικά νησιά στην περιοχή του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου. Το ελεκτικό συνέδριο υπήρξε απορριπτικό ω προ την κατασκευή τη Μαρίνα, διότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα προέβλεπε την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την προσέλκυση πηγών εσόδων εκτό του τουρισμού. Θεωρώ ότι η άποψη αυτή είναι περιοριστική και δεν λαμβάνει υπόψη τη τι ιδιαιτερότητε τη νησιωτικότητα. Σα μιλώ και σαν νησιώτη που έχω βιώσει τι δυσκολίε, τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα μια νησιωτική περιοχή σε σχέση με μια υπηρετική οι μαρίνε, εκτό των πολυτελών σκαφών, φιλοξενούν βάρκε ψαράδων και μικρά πλοιάρια, με τα οποία διευκολύνεται η διασύνδεση των πολιτών που διαμένουν σε κοντινά νησιά. Η αντίρρηση τη Επιτροπή συνίσταται στο ότι το έργο υλοποιήθηκε βάσει προγράμματο με τον επιχειρησιακό στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη κόμβων μεταφορών, επικοινωνία και εύκολη πρόσβαση στα νησιά και με την οποία συμφωνώ. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, αλλά και άλλες οι οποίες έχουν πολλά και μικρά νησιά, η βελτίωση της διασύνδεσης με την υπηρετική χώρα έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για τις νησιωτικές περιοχές το ζητούμενο δεν είναι μόνο η σύνδεσή τους με τα υπηρετικά της χώρας, αλλά και η ύπαρξη επαρκών διασυνδέσεων μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται ενδονησιωτικοί κόμβοι μεταφορών και προωθείται καλύτερα η κινητικότητα των πολιτών αλλά και εμπορικέ συναλλαγές. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Σταυρακάκη και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σκυλακάκη. Αυτή η έκθεση είναι πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ένα, κρούει το κουδόνα του κινδύνου. Τα χρήματα που δαπανούμε σε υποδομές δεν δαπανούνται με σωστό τρόπο. Τώρα η Κομισιόν βάζει τα δυνατά της ε, κατά την παρουσίαση αυτού του θέματος, αλλά το να ε, ε, κατασκευάζουμε λιμάνια τα οποία όμως μετά από 2, 3, 4 χρόνια δεν, δεν λειτουργούν, δεν έχουν συνδέσεις κλπ. Δεν είναι σωστή διαχείριση, είναι λάθος διαχείριση. Η έκθεση δεν πηγαίνει παραπέρα Δηλαδή, ποια είναι τα ποσοστά χρησιμοποίηση, ποια είναι τα οικονομικά ωφέλη που παρέχουν τα λιμάνια. Δεν μπαίνουμε σε μια οικονομική ανάλυση αναφορικά με τις επιπτώσεις των λιμανιών στις περιοχές και το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Αυτοί είναι θεμελιώδεις κανόνες εάν τα κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο, φανταστείτε τι θα προκύψει αν κάνουμε μια περισσότερο σε βάθος μελέτη και εξέταση. Έχουμε δει τι συμβαίνει και θα πρέπει να μπούμε πιο βαθιά για να δούμε πώς ακριβώς δαπάνουν τα χρήματα. Πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κοινωτικών πόρων. Ζούμε μια οικονομική κρίση. Παντού γίνονται περικοπές. Και θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο πανάμε τα χρήματα. Υπάρχουν ζητήματα τα όπου το συνέδριο βλέπει τα πράγματα <clears throat> λίγο πιο γραφειοκρατικά. Άνθρωποι που φτάνουν στα νησιά με πλοία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μαρίνες ε, για να κυκλοφορήσουν, να μετακινηθούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι, ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι τα αποτελέσματα για τις τοπικές οικονομίες. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για το πρώτο ερώτημα, νομίζω ότι έδωσα κάποια στοιχεία. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι από τα τέσσερα ανολοκλήρωτα προγράμματα κατά τη, διά... κατά τη στιγμή του ελέγχου, ένα μόνο δεν ολοκληρώθηκε λόγω νομικών και διοικητικών προβλημάτων. Στο Πρίντεζι, στο νότο της Ιταλίας. Για το δεύτερο ερώτημα, όσον αφορά τη Μαρίνα στην Ελλάδα, συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Σταυρακάκη ότι το θέμα δεν είναι δηλαδή ότι η Μαρίνα δεν, είναι, δεν συνάδει με τους στόχους υποδομής μεταφορών. Το θέμα είναι κατά πόσο συμμετέχει αυτό στους στόχους τοπικής ανάπτυξης και κατά πόσο ε, δημιουργεί οικονομικά ωφέλη για την περιοχή. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και αυτό ε, συνάδει με τους στόχους της πολιτικής συνοχής δεν υποστηρίζουμε υποδομές απλώς και μόνο επειδή συμφωνεί με την ε, ε, πολιτική μεταφορών ή με άλλες τομεακές πολιτικές, αλλά θέλουμε να δούμε κατά πόσο συμμετέχει πράγματι στην ίδια την περιφερειακή ανάπτυξη. Για το τρίτο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το προηγούμενο βέβαια, ε, το ερώτημα της αποτελεσματικότητας είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε κατά πόσο αυτή η υποδομή δημιουργεί τα οικονομικά ωφέλη που προσδοκούμε. ειδικότερα όταν πρόκειται για ε, δημόσια χρηματοδότηση. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ε, ε, περίπτωση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας που δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια. Γι' αυτό δίνουμε τώρα μεγαλύτερη προσοχή στην απόδοση, στα αποτελέσματα και ειδικότερα ε, εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου που έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης ε, της απόδοσης και παρακολούθησης απόδοσης ε, σε τακτική βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει κάποια ερώτηση που να εκρεμεί προς το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, θέλετε μήπως να λάβετε το λόγο για ερωτήσεις που να σας αφορούν ή να κλείσουμε καλύτερα το θέμα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι πολύ σημαντικές οι θαλάσσιες μεταφορές Ε, υπάρχει το πρόγραμμα Μαρκοπόλο το οποίο σχεδιάστηκε μεταξύ άλλων για να μεταφερθούν οι οδικές μεταφορές σε άλλα μέσα μεταφοράς. Επίσης, εξετάζουμε την εσωτερική ναυσιπλοεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, για την έκθεση αυτή σήμερα και είτε εγώ είτε κάποιος από τους ε, συναδέλφους μου που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο αυτού του θέματος ε, θα επανέλθουν στο εγγύς μέλλον ε, για να συζητηθούν και άλλες εκθέσεις τις οποίες και σας ανέφερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συγητής, επιθυμείτε κύριε συγητά να λάβετε το λόγο. Θέλετε να κλείσετε το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Σχετικά με την έκθεσή μου, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια που άκουσα. Αυτό που έχω να πω είναι το εξή. Ε, ναι, όντω αποτελεί ένα να κινδύνου σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σίγουρα θα έχουμε τις νέες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική. κατά πόσον θα ε, θα ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο θα έλεγα αν θα συνεργάμε κάποια συμπεράσματα τόσο εμείς όσο και η Κομισιόν αυτή είναι οι παλιές χώρες όπως η Ιταλία παραδείγματος χάρη που αντιμετωπίζουν προβλήματα και παρατηρούμε ότι οι κυβερνήσεις ε, μεγάλων χωρών ε, κάνουν τα στραβά μάτια στις εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, τον εισηγητή και την ε, Επιτροπή για την απάντηση, τις απαντήσεις που έδωσε αυτά τα θέματα. Πάμε τώρα στο επόμενο και τελευταίο ε, θέμα για σήμερα πριν από τις συνεδρίες των συντονιστών. Πρόκειται για την ειδική έκθεση σχετικά με την Eurostat. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να καλωσορίσω ως ε, εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου τον κύριο Λουί Γκαλία. Ο εισηγητής μας είναι ο Τάμας Ντότζ. Τάμας, ε, θέλετε να λάβετε το λόγο, παρακαλώ, ε, για να μας κάνετε τις αγωγικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πολύ σύντομα είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια. ενώπιον του εκπροσώπου του ελεγκτικού συνεδρίου του κυρίου Γκαλέα και της Eurostat. Θα ήθελα να πω καταρχάς το εξής, ότι το να μιλάει κανείς για στατιστικές είναι περίεργο. Όλοι ξέρουμε ότι για τις στατιστικές μόνο ηρωνικά αστεία μπορούν να γίνουν. Ότι υπάρχουν τρεις τρόποι να πει κανείς ψέματα, να καλύψει την ασφάλεια, να πει κάτι το οποίο δεν ισχύει ή τέλος πάντων να χρησιμοποιήσει στατιστικές. Σε ορισμένες δικτατορίες μάλιστα η πολιτική ηγεσία λένε πίστευαν σε στατιστικές ε, που είτε παραποίησαν είτε τις δημιούργησαν οι ίδιες οι δικτατορίες. Εν ολίγες τέλος πάντων σπάνια λέμε καλά πράγματα για τη στατιστική παρά το γεγονός ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Και κυρίως ε, γιατί ε, της, ε, στα τελευταία, τα τελευταία δέκα χρόνια φάνηκε σε πολλά κρατημέλη ότι στατιστικά δεδομένα είτε είχαν παραποιηθεί είτε δεν ευθυγραμμίζονταν ε, δεν, δεν αντανακλούσαν την πραγματικότητα ούτε αντανακλούσαν την οικονομική κατάσταση στην εν λόγω χώρα από την οποία προέρχονταν. Πέρα βέβαια από το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ανταπόκριση ε, στην οικονομική κρίση μας έδειξε ότι η στατιστική έχει ένα ρόλο και κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού εξαμήνου και οι δείκτες της οικονομικής κατάστασης μας δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή Χρειαζόμαστε λοιπόν τα πιο ακριβή στατιστικά δεδομένα. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα γι' αυτό ακριβώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Γκαλέα και στους συνεργάτες του για την ε, πολύ διεξοδική δουλειά τους. Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που αναφέρω στην έκθεσή μου. Μπορώ να σας πω εν ολίγης ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγησή σας, την οποία δημοσιεύσατε στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στον τίτλο της ειδική έκθεσης, το ερώτημα είναι, το ερώτημα απαντάτε εντός της έκθεσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurostat μπορούν να συνεισφέρουν στην παραγωγή αξιόπιστων και σωστών στατιστικών ε, στοιχείων. Όμως έχουμε πάρα πολλή δουλειά, για να το πω ευγενικά, ακόμη για να το πετύχουμε αυτό. Γιατί το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα, ε, σύστημα, χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση. Μιλάω και για τις προδιαγραφές και για τις ευρωπαϊκές στατιστικές καμπύλες ε, που δείχνουν τη λειτουργία του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν είναι δεσμευτικοί. Η Eurostat σε ένα βαθμό δεν μπορούσε καν να, να, να εφαρμόσει τους κανόνες που αναφέρονταν ε, σε σχέση με την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων και σε ορισμένα υπάρχει μεγάλη απόκληση από το σύνολο των προδιαγραφών που είχαν συμφωνηθεί. Κατά την αξιολόγησή μου λοιπόν, φαίνεται και από τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια δουλειά, την αρχή μιας δουλειάς αναθεώρησης του ε, συστήματος. Ένα νέο σύνολο κανόνων ε, συζητά τώρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα και αυτό είναι το τρίτο τμήμα της εκθεσής μου που εστιάζει στις ειδικέ συστάσεις. Με πολύ χαρά θα ακούσω τις συστάσεις σας. Μπορώ να σας πω ότι τρία ουσιαστικά θέματα χρήζουν συζήτησης Πρώτον, κατά πόσο οι αλλαγές είναι επαρκείς, οι αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την άποψή μου, ως εισηγητή, όχι είναι η απάντηση. Οι συστάσεις πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Δεύτερον, κατά πόσο η, η εκλογή του διευθυντή της Eurostat εξασφαλίζει τους σωστούς κανόνες για την ανεξαρτησία της Eurostat. Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και να τονίσω εδώ ότι το επταετές πλαίσιο προϋπολογισμού που θα τεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δείχνει σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης. Ε, η Eurostat έχει πολύ μεγαλύτερο άχθος εργασίας ε, και ο προϋπολογισμός δεν έχει ευθυγραμμιστεί με την αύξηση αυτού αυτής της δουλειάς που πρέπει να κάνει η Eurostat για να μπορέσει να, οδηγη, να, ε, να οδηγηθεί στην παραγωγή σωστών και αξιόπιστων στατιστικών. Και τρίτο πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι το καθεστώς ε, του, της συμβουλευτικής ομάδας, του ε, Συμβουλευτικού ε, Συμβουλίου των Στατιστικών, που να έχει αρμοδιότητες που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της Eurostat, και μεγαλύτερος έλεγχος και καλύτερος έλεγχος των ευρωπαϊκών στατιστικών. Χαίρομαι, ε, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η έκθεση αυτή του ελεκτικού συνεδρίου. Ελπίζω να ληφθεί υπόψη ε, στη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στατιστικών, το οποίο πρέπει να βελτιωθεί και να τροποποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστούμε και εμεί τον εισηγητή και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή του ελεγκτικού συνεδρίου να τοποθετηθεί και αυτό ο κύριο Καλία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Deutsch, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτή την ακρόαση σχετικά με την ε, ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που σε αυτή την περίπτωση εξετάζει δύο βασικά θέματα που αφορούν στη Eurostat. Το πρώτο θέμα είναι ο Ευρωπαϊκός Στατιστικός ε, Κώδικας και το δεύτερο που εξετάζεται είναι η απόδοση της Eurostat κατά την ε, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος. Το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ντόιτς, ε, του εισηγητού, συνοψίζει πάρα πολύ καλά τα πορίσματα του συνεδρίου και παραπέμπει στα κρίσιμα θέματα και έτσι λοιπόν και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος στην παρέμβασή μου. Τρία θέματα θέλω να αναφέρω. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί τον πρακτικό κώδικα της Eurostat ως ένα ε, προαπαιτούμενο για να υπάρχει εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα. Το συμπέρασμά μας είναι ότι δεν εφαρμόζεται πλήρως ακόμα ο κώδικας. Έτσι λοιπόν ε, προέκυψαν δύο βασικά απορίσματα σε σχέση με την ε, προσήλωση στον κώδικα. Σήμερα αυτό το θέμα ε, είναι θέμα αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη ανάμεσα στη Eurostat και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Τα συστήματα της ε, επαλήθευσης εξακολουθούν να είναι αρκετά αδύναμα. Και όσον αφορά στο ποιος ευθύνεται για την εφαρμογή του κώδικα, εμείς παρατηρήσαμε ότι η εφαρμογή του κώδικα εξαρτάται εν μέρη όχι μόνο από τη Eurostat και από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, αλλά εξαρτάται και από τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες ε, καλούνται να ε, εισάγουν μεταρρυθμίσεις και να υιοθετήσουν ε, τις δικές μας τις προδιαγραφές. Ως έχουν τώρα τα πράγματα, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες πολλές φορές δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ποιότητα των δεδομένων και όλα τα άλλα που προβλέπει ο κώδικας. Το συμπέρασμά μας λοιπόν είναι ότι όλα αυτά προκύπτουν από μία ε, συγκαλυμμένη αμφισημία ως προς τον κώδικα. Για μας, ε, για τον, σχετικά με τον κώδικα, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό το γιατί ορισμένες αρχές του κώδικα ε, δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Όσον αφορά το δεύτερο ε, στοιχείο της έκθεσής μας, δηλαδή την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος 2008-2012, ε, το συνέδριο συνεπέρανε ότι η Eurostat δεν έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα αυτό ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου και λογοδοσίας. Διαπιστώσαμε ότι πρέπει να υπάρξει νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Το νέο στατιστικό πρόγραμμα μέχρι το 2014 πρέπει να ομολογήσουμε εξετάζει τα απορίσματα του συνεδρίου και προσφέρει καλύτερη η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων προσφέρει και νέες μεθόδους για τη συγκέντρωση ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων. Βεβαίως θα δούμε πώς όλα αυτά θα υλοποιηθούν κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Τέλος, ε, τα ε, συμπεράσματα είναι κάτω από τρεις επικεφαλίδες. Πρώτον, τα πολύ γενικά. Εμείς πιστεύουμε ότι ευρωπαϊκά αξιόπιστα και ε, αξιόπιστα δεδομένα, αυτό είναι ε, κοινή ευθύνη. Πρέπει να υπάρξουν σοβαρές δράσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλυθούν και από την Κομισιόν και από τα κρατη και από τις στατιστικές υπηρεσίε. Όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα. Ε, η δεύτερη δέσμη συστάσεων αφορά στην πλήρη εφαρμογή του κώδικα πρακτικής εγώ ε, δεν θέλω να ε, πω τίποτα πιο πολύ, γιατί ε, αναφέρονται όλα αυτά στις συστάσεις. Και η τρίτη δέσμη συστάσεων αφορά το στατιστικό πρόγραμμα. Εδώ το εμείς επισημαίνουμε προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές και από την Κομισιόν για το μέλλον. Και τέλος θέλω να προσθέσω ότι η Επιτροπή και η Eurostat έχουν ήδη λάβει μέτρα σε σχέση με την έκθεσή μας και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς πιστεύουμε ότι ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά και η Eurostat πρέπει να δεχθεί τις συστάσεις ε, του συνεδρίου έτσι ώστε να υπάρχει συστηματική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη φάση εφαρμογής ε, του νέου Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος για τα έτη 13 έως 17. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ja, vielen Dank für die Kommission. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους της Επιτροπής ε, καλωσορίζω τον κύριο Έβερας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσάς να τοποθετηθείτε ή μήπως ε, θέλετε να απαντήσετε μόνο σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, μου δίνετε το λόγο και μου δίνετε και τη δυνατότητα να πω ορισμένα πράγματα κατά τη συζήτηση αυτή. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα, όπω επίση και το Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί εξετά... έκαναν αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση για το ρόλο των στατιστικών και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για τις έγκυρες και αξιόπιστες στατιστικές και την... Ε, τα στατιστικά στοιχεία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Το θέμα των έγκυρων στατιστικών αναφέρθηκε ήδη πολλές φορές, είχε αναφερθεί πολλέ φορέ και είναι σαφέ ότι για όλους μας ε, είναι εξίσου σαφές ότι οι στατιστικές είναι σημαντικό τμήμα της ε, ευρωπαϊκής υποδομής. Ε, οι αποφάσεις που βασίζονται στην πολιτική χρειάζονται υψηλού επίπεδου στατιστικέ προκειμένου να ληφθούν. Εκτιμούμε τις ε, συστάσεις ε, του ελεγκτικού ε, συνεδρίου, όπως και τον τρόπο με τον οποίο τις έχει μεταγράψει σε έκθεση ο εισηγητής κ. Ντόιτς, γιατί νομίζω ότι αντανακλούν πολύ σωστά τα βήματα που θέλαμε να ακολουθήσουμε πριν από ένα-δύο χρόνια. Η Eurostat λοιπόν συμφωνεί σχεδόν με όλες τις συστάσεις του εισηγητή στην έκθεσή του της 19 η Δεκεμβρίου του 2012. Το σχέδιο δράση στο οποίο ανέφερε και ο κύριος Γκαλέα να φέρει τα στοιχεία που έχουν ήδη δρομο, τη στρατηγική που έχει ήδη δρομολογηθεί, που πρόκειται να δρομολογηθεί. Οι, οι συγκεκριμένες συστάσεις είναι πάρα πολύ ε, σύντομες, συγκεκριμένες και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα τις μεταφράσουμε σε πράξη γιατί οι συστάσεις αυτές μοιάζουν, πάρα πολύ, ε, σε μεγάλο βαθμό με τις συστάσεις του εισηγητή, του κυρίου Ντόιτς. Θα ήθελα να τονίσω μερικά στοιχεία. Πρώτον, ο ρόλος που τον ανέφερε και ο κύριος Γκαλέα, του κώδικα ε, πρακτικής. Ο κύριος Ντόιτς το ανέφερε αυτό. Αυτός ο κώδικας αναπτύχθηκε το 2007 στο πλαίσιο του συστήματος αυτορύθμισης και βελτιώνεται συνεχώς, εστιάζει όλο και περισσότερο ε, στο Συμβουλευτικό ε, Συμβούλιο των, ε, του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, ε, κάτι το οποίο επίσης είπε ο κύριος Γκαλέν να μην βλέπουμε μόνο τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ή τους παροχή στατιστικών, αλλά να δούμε και το ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κώδικας πρακτικής, και το λέω αυτό σε σχέση με τη δέσμευση των κυβερνήσεων για την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου στατιστικών, μέσω διευκόλυνσης της παρακολούθησης καθ' όλη τη... στο πνεύμα του κώδικα πρακτικής. Είναι πολύ σημαντικά θέματα, γι' αυτό Ευχαριστούμε πολύ το Κοινοβούλιο ε, για την προσπάθειά του να πείσει τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις ότι είναι και το περιβάλλον εντός του οποίο δουλεύουν πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου για να υποστηρίζουν ε, την παραγωγή στατιστικών ε, να πω επίσης ε, ότι η ίδια η Eurostat ε, ανανέωσε τη δεσμευτή στις 17 Δεκεμβρίου ε, για το θέμα της εμπιστοσύνης και της ανεξαρτησίας της. Ένα ακόμη θέμα που αναφέρθηκε είναι το κομμάτι του προϋπολογισμού και χάρηκα που ο κύριος Ντόιτς το ανέφερε γιατί είναι κάτι το οποίο ε, στο πλαίσιο της ε, τρέχουσας ε, κατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τόνισα ήδη ότι οι στατιστικές είναι μία από τις βασικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπ' αυτήν την έννοια η παραγωγή τους πρέπει να εξασφαλίζεται. Και το λέω αυτό σε σχέση με τα θέματα του προϋπολογισμού. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις στο σχέδιο έκθεσης αλλά και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου με τις, ε, για τα οποία έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Ε, ένα από αυτά είναι ο ρόλος της ΕΣΓΑΠ. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα θεωρημένο ρόλο ο, ε, πιο ανεξάρτητο της ΕΣΓΑΠ, αλλά πρέπει να βλέπουμε και την αξιολόγηση ομοτήμων στον κώδικα της πρακτικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της ε, εντολής που έχει ληφθεί βάση της νομικής βάσης, ε, πρέπει κάποιος να εποπτεύει τις επαληθεύσεις ε, και αναφέρομαι και ε, στην ε, Συμβουλευτική Επιτροπή της Όλαφ ε, στην απόφαση, στην δέσμευση που αναλάβαμε στις 17 Δεκεμβρίου αναφερθήκαμε ειδικότερα στην ανεξαρτησία και διευκρινίζει γενικώς ειδικώς το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής μεταξύ άλλων έχει ανανεώσει τη δέσμευτή του για την παραγωγή σωστών στατιστικών. Η ΕΣΚΑΠ είναι ένα τεχνικό σώμα που ελέγχει την αξιολόγηση ομοτύπων και έρχεται σε επαφή με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς και τα κράτη-μέλη. Έχω και κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το ρόλο της ΕΣΓΑΠ. για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας ε, της Eurostat ε, μιλώ. Βάσει του κανονισμού 23 έχουμε παρκή εξουσία για το πλαίσιο, στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας επιλογής. Το θέμα τώρα βέβαια είναι η εστίαση στους κανόνες των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών των γενικών διευθυντών των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών, που είναι η Εθνική Αρχή Στατιστικών, που πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχει έναν εποπτικό ρόλο όλων των υπολέπων φορέων που συμμετέχουν στην παραγωγή επισήμων στατιστικών. Πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και σωστή παρακολούθηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Ντόιτς και τον Ελεκτικό Συνέδριο για τις εκθέσεις τους ε, που με τις δύο εξαιρέσεις που ανέφερα με ικανοποιούν ιδιαιτέρως και τις ευχαριστώ πολύ για αυτές. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα έχει το λόγο η συνάδελφός μας. Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις επιβεβαίωσαν ότι τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία ε, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Χρησιμοποιούνται από όλους τους τομείς, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την ε, εξέταση της αποτελεσματικότητας ε, ό,τι φορά την χρήση αυτών των κονδυλίων. Όλο και οι περισσότερες αποφάσεις εξαρτώνται από αυτές τις στατιστικές. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το ότι υπάρχουν αυτά τα σχόλια από πλευράς ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. γεγονό είναι ότι λείπουν κάποια μέτσα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Ε, πιστώνω ότι η Eurostat ε, και τα κράτη-μέλη φέρουν μια κοινή ευθύνη για την τήρηση της ε, εμπιστευτικότητας και της αποτελεσματικότητας ε, των στατιστικών. Θα πρέπει το σύστημά μας να στηρίζεται όχι μόνο στην ενίσχυση της ε, ανεξαρτησίας των στατιστικών υπηρεσιών αλλά και την ανεξαρτησία των επικεφαλής των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Ε, οι οποίες στατικές υπηρεσίες πρέπει να παίρνουν εντολές και οδηγίες από τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό το λόγο προτείνω προτροπολογίες που πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη είναι η συνάδελφος κυρία Αντρέασεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να διευκρινίσω κάποια ζητήματα που έθιξε ο εισηγητής σε σχέση με το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Από ό,τι κατάλαβα, ο εισηγητής είπε ότι ο κώδικας δεοντολογίας δεν ήταν ικανοποιητικός. Ενώ το ελεγκτικό συνέδριο δήλωσε ότι δεν εφαρμόστηκε ορθά. Αυτά είναι δύο διαφορετικά προβλήματα. Τι από τα δύο συμβαίνει. Είναι ικανοποιητικό ή όχι και εφαρμόζεται ή όχι. Η το της ε, καταστάσεως την οποία ανέφερε ο συνάδελφος σχετικά με την οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανησυχητικό να λαμβάνουμε γνώμη του συνεδρίου να λέει ότι το σύστημα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μάθει το μάθημά μας, διότι κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί. Άρα είναι εκπληκτικό να έχουμε περάσει εκτός της αμοιβαίας εμπιστοσύνη, να την έχουμε ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο και να μην μιλήσουν για, μίλησαν για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας. Η Κομισιόν μίλησε για κοινή ευθύνη Ίσως να υπάρχει κοινή ευθύνη, αλλά κάποιος θα πρέπει να ηγείται, να είναι επικεφαλής. Οι ε, υπηρεσίες, ε, ε, εθνικές υπηρεσίες στατιστικής και οι κυβερνήσεις φέρουν ευθύνη. Αλλά η Eurostat θα πρέπει να ηγηθεί. Διαφορετικά, τι λόγο ύπαρξη έχει. Μόνο και μόνο για να συλλέγει τις στατιστικές πρόσθετα από τα κράτη-μέλη, όχι θα πρέπει να εξετάζει την ποιότητα των στατιστικών αυτών και ότι ο κώδικας διοντολογίας εφαρμόζεται. Η ερώτησή μου είναι προς την Κομισιόν. Δέχονται τον ε, ηγετικό ρόλο της ε, Eurostat. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κάποιος άλλος λόγο. Α, όχι, κυρία Κρέσλε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα για μένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτή είναι μια ερώτηση προς την Eurostat. Είναι σημαντικό ε, οι απάτες που έγιναν στα ελληνικά στατιστικά δεδομένα να μην επανέλθουν. Πρόεδρος, ε, θα ήθελα λοιπόν τώρα να ζητήσω από την Επιτροπή καταρχήν να απαντήσει ή αν θέλετε από τον εκπρόσωπο της Eurostat, δεν ξέρω ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Κοιτάξτε, θα ήθελα να απαντήσω πρώτα στην ερώτηση της κυρίας Ανδρέασεν. Ο κώδικας πρακτικής προέκυψε σε ένα ρυθμιστικό σύστημα και ελέγχεται από ε, μελέτες και έρευνες ομολόγων, ο ομοτήμων αν θέλετε, αυτό είναι ένα από τα θέματα ε, που αφορά στα αυτορυθμιστικά συστήματα. Έχουμε διαπιστώσει τις αδυναμίες του συστήματος και νομίζω αυτές επισημάνθηκαν και από το ελεγκτικό συνέδριο. Γι' αυτό λοιπόν επιφέραμε διάφορες αλλαγές. Η μία εξ αυτών που αναφέρθηκε είναι η ιδέα για τη δέσμευση ως προς την εμπιστοσύνη. να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη όπως είπε η κυρία Αντρέασεν. Αυτό θα αλλάξει. Η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους θα υπογράφει και θα αγκιάται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων. Άρα δηλαδή η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα μεταφέρεται σε ένα σύστημα με σαφείς ε, υπογραφές ε, για ανάληψη υποχρεώσεων. Η κοινή ευθύνη και αυτή έχει σχέση με όλα αυτά. Είναι σαφές ότι η Eurostat παίζει εδώ πρωταρχικό ρόλο. Εμείς καθορίζουμε την αναθεώρηση που λαμβάνει η χώρα. Έχουμε δείξει στα κράτη-μέλη ε, το πώς μπορεί να εφαρμοστεί μια δέσμευση για την ύπαρξη εμπιστοσύνη και προσπαθούμε να ε, πείσουμε την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τη σημασία της ε, δέσμευσης ε, ε, που καθιστά σαφές ότι θα υπάρχει κοινή ανάληψη ευθυνών υπό την καθοδήγηση της Eurostat. Ο κανονισμός 223 είναι πολύ σημαντικός και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στα ομάδα εργασία του Συμβουλίου έχουν ήδη ε, προσκληθεί επανειλημμένα να συνεργαστούν σε ομάδες εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Γκρέσλε, βεβαίω είναι ένα ερώτημα ή μία παρατήρηση που με οδηγεί στο να πω ότι πέρυσι προβλέφτηκαν πολλά εργαλεία που πλέον διασφαλίζουν ότι δεν θα επαναληφθούν ελληνικής ε, φύσεως σε στατιστικά δεδομένα. Βεβαίως η ζωή είναι δύσκολη και περίπλοκη. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και προσπαθούμε, όπως σας είπα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εγγυηθούμε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Έχουμε το συμβουλευτικό όργανο ε, των Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δομένων. Έχουμε την ECC ε, Επιτροπή, αναθεωρήσαμε τον κανονισμό, τον νέο κανονισμό 223, την απόφαση για τη Eurostat. Έχουμε διάφορους ε, κανονισμούς για τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονται τα στατιστικά δεδομένα. Εδώ και πολλά χρόνια οι κανονισμοί μας εστιάζονται σε θέματα ποιότητας και ποιοτικών εκθέσεων. Θα μπορούσα να συνεχίσω ώρες ολόκληρες για να σας ενημερώσω για το τι έχουμε κάνει. Βεβαίως ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ εγγύηση 100% αλλά εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία για να ε, εμποδίσουμε τέτοιου είδους ε, φαινόμενα. Όσον αφορά στην επόμενη ερώτηση, νομίζω ότι στην απάντηση προς την κυρία Αντρέασεν απάντησα στον κανονισμό σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς όπως τον ε, καταρτίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκαλέα από το Ελληνικό Συνέδριο. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθησαν από τους ευρωβουλευτές. Εξακολουθούμε να είμαστε της απόψεως ότι χρειάζεται μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών, για σεβασμό όλων των αρχών του κώδικα, δεύτερον διαφανέστερη και πιο ανεξάρτητα διοριστήσα ε, επιτροπή, επίσης ε, ανεξαρτησία, εποπτεία και εφαρμογή των κανόνων ε, θα οδηγηθεί θα οδηγήσει σε μια αποτελεσματικότερη Eurostat ε, και θα είναι και πιο χρήσιμη για τους πολίτες και μιλάω σε σχέση με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των στατιστικών. Η Επιτροπή Εμπιστοσύνης είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είμαστε ακόμη πεπισμένοι ότι μπορεί να υποκαταστήσει ενός, ένα μηχανισμό ε, ισχυρό επαλήθευσης και ανεξάρτητο. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γκαλέα, γιατί πραγματικά τα συνόψισε όλα πολύ σωστά, οπότε τρία θέματα θα ήθελα να θέσω εγώ. Πρώτον, να τονίσω ότι το ερώτημα που έθεσε ο, το ζήτημα που έθεσε ο εκπρόσωπος της Eurostat Μπορούμε να μιλούμε για ανεξαρτησία μόνο αν έχουμε τις απαραίτη, τους απαραίτητους πόρους στον προπολογισμό για την πραγμάτωση αυτής της ανεξαρτησίας. Για την ώρα πως έχουν όμως τα πράγματα, οι πόροι για τη λειτουργία της Eurostat, τέλος πάντων τμήμα των πόρων της, φτάνουν στη Eurostat μέσω διαφορετικών γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής. Θα ήταν πολύ καλύτερο οι πόροι αυτοί να βρίσκονται σε μια γραμμή του προϋπολογισμού, ειδικά για τη Eurostat. Στα επόμενα 7 χρόνια η Eurostat θα έχει πολύ περισσότερα καθήκοντα και για να μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντα αυτά, ανεξάρτητες αντικειμενικές στατιστικές είναι απαραίτητες γιατί είναι το βασικό υλικό αποφάσεων για τις αποφάσεις. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δύο βασικά ε, σημεία υπάρχουν στην έκθεσή μου με τα οποία διαφωνεί σημεία 7 και 13 και έχουν να κάνουν με την ΕΣΓΑΜ και το διορισμό ή την αποπομπή των διευθυντών των στατιστικών υπηρεσιών. Εξακολουθώ να επιμένω όμως στη θέση μου. Και το τελευταίο ερώτημα που έθεσε η κυρία Σεν, στο οποίο απαντώ τώρα, είναι ότι το περιεχόμενο του κώδικα πρακτικής ήδη είναι κάπως προβληματικό και η εφαρμογή του είναι επίσης προβληματική. Τότε, άρα και το περιεχόμενο και η εφαρμογή παρουσιάζουν προβλήματα Τα προβλήματα αυτά μπορούν να επιληθούν βάσει του άρθρου 233. Είναι και καινή ώρα νομίζω να αποφασίσουμε πώς ε, η λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμορφώνεται πιο πολύ προς τους κανόνες. Εγώ δεν βλέπω πραγματικά κανένα επιχείρημα που να αντίκειται σε αυτό το στατιστικό σύστημα που θα εκπροσωπεί όντως τα καθήκοντα της Eurostat. Αν έχουμε μία ενιαία ε, μεθοδολογία και ενιαίες προδιαγραφές, τότε αυτό το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα μπορεί να λειτουργήσει. Συνοψίζοντας, να σας ευχαριστήσω όλους για τα πολύτιμα σχόλιά σας και το ελεγκτικό συνέδριο για τη γνωμοδότησή του. Αναμένω εναγωνίως τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, κύριο Γκαλία από το ελεγκτικό συνέδριο και τον κ. Πιτευκάς, αν ε, πρόφερα σωστά τα ονόματά σας. Και ε, ευχαριστώ και την Επιτροπή που συμμετείχε στη συζήτηση. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και έτσι λοιπόν κλείνει η επίσημη συνεδρίαση, ε, η ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής μας και Τώρα θα περάσουμε ευθύ αμέσω στι συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση των συντονιστών.